Uh, dear colleagues, could the meeting? Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε πάλι τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω όσους βρίσκονται εδώ στην αίθουσα για το επόμενο τμήμα της συνεδρίασης ΑΦΚΟ. Να σας ενημερώσω ότι ήδη από την πρώτη μέρα αυτή της θητεία ε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ασχολείται, προσπαθεί να εντοπίσει πράγματα που δεν λειτουργούν ε, στην Ευρώπη για να βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τις πολιτικές της, χρησιμοποιώντας ε, τα μέσα που μας δίνει η ισχύουσα συνθήκη. Πιστεύουμε όμως επίσης ότι πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από την ισχύουσα συνθήκη, να κοιτάξουμε το μέλλον, να δούμε πώς μπορούμε περαιτέρω να βελτιώσουμε τον τρόπο που η Ευρώπη αποκρίνεται στους ε, πολίτες της, ε, στις ε, ανάγκες ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, δημοκρατία και την ε, λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το τοπικό, το εθνικό, το περιφερειακό. Έτσι, αναπτύξαμε ένα ενδιαφέρον για τι θεσμικές προσαρμογές ε, στη μερωτική ανάπτυξη της Ένωσης. Εξετάζουμε λοιπόν το μέλλον, κυρίως όσον αφορά την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον τρόπο που έχει δομηθεί, τον τρόπο που λειτουργεί, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν εξετάζουμε τις επιμέρους πολιτικές ε, αυτές έχουν να κάνουν με μια άλλη μεγάλη πρόκληση. Πώς η Ευρώπη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο των πολιτικών της ε, για να ε, αποδίδει πιο αποτελεσματικά. Και έτσι φτάνουμε στη σημερινή συνεδρίαση, διότι ε, βρισκόμαστε στην τελική φάση των εργασιών για δύο εκθέσεις που συζητήσαμε και πριν ένα χρόνο μαζί σας. Βρίσκονται λοιπόν τώρα στο τελικό στάδιο και στις 8 ε, Δεκεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ελπίζουμε στις αρχές Φεβρουαρίου να αποτελέσουν ε, την ε, βάση για συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει το μέλλον και τις αλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπα και το πρωί, διαμορφώνουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα λάβουμε όμως και την ε, Λευκή Βίβλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και ελπίζουμε να δούμε και την εφαρμογή της, ε, του οδικού χάρτη της Μπρατισλάβα που περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές. και ελπίζουμε επίσης ότι θα έχουμε μια καλή συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων ώστε να έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε το περιεχόμενο των εκθέσεών μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με εισαγωγή από δύο πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες. Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον καθηγητή Μάριο Μόντι, που επίσης ε, διατέλεσε επίτροπος δύο φορές. Και έχουμε μαζί μας και τον Αντώνιο Βιτορίνο, που επίσης ε, διατέλεσε επίτροπος δικαιοσύνης και εσωτερικών ε, υποθέσεων. Ε, ήταν όμως επίσης πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ε, Υπουργός ε, Αμήνης και Πρόεδρος του Ταγματικού Δικαστηρίου. Ε, έτσι έχει ζωή, όλα μεγαλώνουν τα βιογραφικά μας. Αντώνιο, θα ήθελα να δώσω πρώτα σε σένα το λόγο. Ε, για να ακούσουμε τι μπορείς να μας πεις ε, για να μας εμπνεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές ε, και αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθώ εδώ σήμερα και να βρεθώ στο ίδιο βήμα με τον Μάριο Μόντι. Πράγματι, επί δεκαετίες ασχολούμαστε με την Ευρώπη και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε και τις επόμενες δεκαετίες του, του πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες και ε, ρεαλιστές. Η παρούσα κρίση που αντιμετωπίζει ε, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν μοιάζει με προηγούμενες κρίσεις. Πάντα λέγαμε εδώ ότι ε, η Ευρώπη θα βγαίνει πιο δυνατή από κάθε κρίση, ενώ νομίζω ότι για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε ε, πιθανή διάλυση της Ευρώπης, πόσο μάλλον ε, μετά από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις ε, υπάρχει μία προϋπόθεση. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η πρόσφατες κρίσεις έχουν οδηγήσει σε διαιρέσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν μόνιμες και να υπονομεύσουν την πολιτική συνένεση μεταξύ των κρατών μελών. Βλέπουμε κάποια δείγματα, κάποιους σχηματισμούς περιφερειακών ομάδων, ο Βοράς κατά του Νότου, η Ανατολή κατά της Δύσης κλπ που μπορεί να είναι αποφασιστικέ για το μέλλον ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ε, τούτου λεχθέντο ε, δεν νομίζω ότι είναι πιθανό πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ να υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξουν οι συνθήκες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στο να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν όσον αφορά ιδιαίτερα τις πολιτικές προτεραιότητες και έχοντας κατά νου ότι οι πολιτικές επιλογές μπορεί να απαιτήσουν θεσμικές προσαρμογές. Καταρχά θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ολοκλήρωση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Συμμερίζομαι τη θέση της ε, καγκελαρίου ε, Άγγελα Μέρκελ που θεωρεί ότι αν το ευρώ αποτύχει διακυβεύεται και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι η βασική μας προτεραιότητα η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, το οποίο σημαίνει δύο πράγματα. Να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στον επιμερισμό του κινδύνου και του ε, επιμερισμού των ευθυνών. Έχουμε λοιπόν την Τραπεζική Ένωση που θα πρέπει να ολοκληρωθεί διότι κατά τη γνώμη μου έχουμε προχωρήσει αρκετά στον έναν τομέα, όχι όμως ε, στον επιμερισμό των κινδύνων. Ε, αναφέρομαι ε, στο Ταμείο Εξυγίανσης των Τραπεζών και στην ε, κοινή εγγύηση καταθέσεων. Στους δύο αυτούς τομείς απομένει ακόμα δουλειά να γίνει και που θα πρέπει να γίνει σύντομα, διότι σίγουρα ε, δεν έχουμε ξεφύγει τελείως από τον κίνδυνο ε, ε, επαναφοράς της κρίσης του ευρώ. Έχουμε λοιπόν ένα εύστραυστο τραπεζικό σύστημα σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν θα σας πω όμως σε ποια. Ο δεύτερος τομέας, κατά τη γνώμη μου, είναι να ξεκινήσουν εις βάθος συζητήσεις του στόχου και της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, διότι αυτό το εργαλείο έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τις ασυμμετρικές κρίσεις βραχυπρόθεσμα. ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα πρέπει να είναι πιο ε, ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας ε, να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα του ευρώ. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αποκλειστικά στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρότι κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει το μέλλον ε, του κοινού μας νομίσματος. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το δεύτερο θέμα είναι να ε, επανέλθουμε στην οικονομική ανάκαμψη και ε, να ξαναβρεθούμε στο δρόμο για τη σύγκληση. Νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές έχουν συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ε, έκθεσή τους που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Εγώ προτείνω μια νέα προσέγγιση να συνδυάσουμε τις διαδικασίες για τις μακροοικονομικές ισορροπίες και την αποτελεσματικότητα των συστάσεων αναχώρα, κυρίως όσον αφορά ε, την ανάγκη για εθνική οικειοποίηση, για αίσθημα ιδιοκτησία όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Κάτι που απαιτεί κατά τη γνώμη μου όχι μόνο αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και αυξημένο ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια τα εθνικά κοινοβούλια μεταφέρουν ε, στην εθνική νομοθεσία τα κεντρικά στοιχεία ε, στα προγράμματα ε, εθνικών μεταρρυθμίσεων. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό σωστά δεν θα υπάρχει αρκετό αίσθημα οικειοποίησης και έτσι θα είναι πιο αποδυναμωμένη η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι αντιμετωπίζουμε διτή πρόκληση. Καταρχάς, θα πρέπει να ε, ξεφύγουμε από την προσέγγιση που έχουμε αυτή τη στιγμή για τις ε, μακροπρόθεσμες ε, ανισορροπίες και να προχωρήσουμε σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα τα οποία να μας επιτρέψουν να επανεξετάσουμε την παραδοσιακή χρήση δαπάνη των διαφορετικών ταμείων. Κατά τη γνώμη μου η παραδοσιακή αυτή η οπτική ε, φτάνει στο τέλος της και εάν θέλουμε να είμαστε πιο προορατικοί ε, για να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει τα διαφορετικά ταμεία και άλλες ε, δυνατότητες χρηματοδότησης και δεν θα πω πολλά για το θέμα αυτό, διότι ξέρω ότι ο Μαριομόντι θα πάρει το λόγο μετά από μένα και έχει πολύ σημαντικό έργο να κάνει ε, βρίσκοντας νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουμε θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε για να προωθήσουμε τις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα. Και για το στόχο αυτό είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, εξετάσει προσεκτικά τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ανάγκη ε, τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup να είναι πολύ πιο προορατικοί κατά την αξιολόγηση του σωρευτικού αποτελέσματος των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Αν δεν έχουμε μεταρρυ... Ε, σωστό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν ε, έχει νόημα ε, να εξετάζουμε ένα-ένα τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα της ε, συνολικής, του συνολικού αντικτύπου τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που απουσιάζει και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πολύ πιο προορατική. Θα κλείσω με μια αναφορά στον θεσμικό αντίκτυπο. Για να είναι πιο αποτελεσματική η διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, πάντα ήμουν υπέρ του να έχει το Eurogroup μόνιμο πρόεδρο. Χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο. Χρειαζόμαστε κάποιον υπεύθυνο που να λογοδοτεί και που να ελέγχεται. Κάποιοι πιστεύουν και μάλλον έχουν δίκιο ότι χωρίς τροποποίηση της συνθήκης Είναι δυνατόν να έχουμε μόνιμο πρόεδρο στο Eurogroup ή ακόμα να δώσουμε την θέση αυτή σε αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Δεν ε, θα μπω τώρα στην νομική συζήτηση το αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Αυτό θα το αφήσω στους εμπειρογνώμονες αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνιμος πρόεδρο του Eurogroup να λογοδοτεί απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα ε, να λογοδοτεί σε ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου αρμόδια για τη ζώνη του ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι και ο βασικός συνομιλητής των εθνικών κοινοβουλίων κατά την ε, συζήτηση των κατευθυντηρίων γραμμών και των βασικών στοιχείων των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης. Δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη για νέους φορείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στο ισχύον πλαίσιο και ιδιαίτερα το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαδικασίε λήψη αποφάσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα ε, όπως είναι η, οικονομική και νομισματική πολιτική είναι πάρα πολύ επαχθής και δεν θα πρέπει να ε, κάνουμε τη διαδικασία αυτή πιο πολύπλοκη, πόσο μάλλον που ε, σε εποχές κρίσης είναι απαραίτητο να λαμβάνονται γρήγορα. Κυρία Πρόεδρε, αυτές είναι οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Θα ήθελα να σας επαναλάβω τις ευχαριστίες μου που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις ε, μπροστά σε ένα τόσο διακεκριμένο κοινό. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Thank you very much. Can I just ask you a question? Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση να σας κάνω, που ίσως πάει λίγο πέραν αυτών που περιμένατε. Διότι αναφερθήκατε στην Ευρωζώνη. Ποιο θεσμικό όργανο πιστεύετε, Αντώνιο, ότι θα έπρεπε να είναι το αρμόδιο για να διασφαλίσει ότι σε αυτή την περίπτωση η Ευρωζώνη θα προχωρήσει περαιτέρω με την ολοκλήρωση και θα διασφαλίσει την ύπαρξη μηχανισμών που θα προστατεύουν την ενιαία αγορά και δεν θα υπονομεύεται αυτό από το γεγονός ότι έχουμε ε, Ευρώπη με χώρες εντός και εκτός Ευρωζώνης και ε, κατά πόσο θα υπάρχει συνέπεια με τις πολιτικές οι οποίες ε, κατευθύνουν την Ευρωζώνη και ε, τους υπολείπους εκτός ευρώ και επίση ε, να αποφύγουμε οποιαδήποτε διάκριση, α την αποκαλέσω έτσι, ε, ε, για τι χώρε εκτό τη Ευρωζώνης. Ποιο θα πρέπει να είναι αρμόδιο για αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ να απαντήσω. Καταρχάς νομίζω ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. παρά το γεγονό ότι έχουμε δύο χώρε που έχουν τη δυνατότητα opt-out και προς, κατά πάσα πιθανότητα σε δύο χρόνια λιγότερο μόνο μια χώρα με opt-out. Όλε οι άλλε θέλουν να τηρήσουν τα κριτήρια και να ενταχθούν στο ενιαίο νόμισμα. Και ε, οι εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά την κοινή πολιτική είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου των Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια κοινή νομοθετική διαδικασία και απομένως έτσι πρέπει να ισχύει. Η νομική εγγύηση της συνοχής του ε, προγράμματος ε, θα πρέπει να αγκιάται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ο νομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών. Όσον αφορά την πολιτική σκοπιά, πιστεύω ότι προκειμένου να αποφύγουμε διακρίσεις και να διασφαλίσουμε πολιτική συνοχή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που θα το διασφαλίσει αυτό. Ήλπιζα ότι θα έλεγατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τέλος πάντων απαντήσατε αυτό που απαντήσατε. Κύριε Μόντι, μήπως θα μπορούσατε να ξεκινήσετε εσείς τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να απευθύνομαι στα μέλη της Επιτροπής σας. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ με το φίλο μου τον Αντώνιο Βιτορίνο. Οι πιθανότητες μας λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα του απομένουν περισσότερες δεκαετίες να δώσει μάχη υπέρ της Ευρώπης από ότι εγώ αλλά τέλος πάντων και εγώ υπό το ίδιο πνεύμα θα μιλήσω. Συμφωνώ και μαζί σας, κυρία Πρόεδρο, και με τον Αντώνιο Βιτερίνο, ως προς το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες της παρούσας συνθήκης και πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο για καλύτερη χρήση της συνθήκης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πω δύο λόγια στο ε, σημείο το οποίο ανέπτυξε ο Αντώνιο Βιτερίνο, κυρίως δηλαδή την οικονομική διακυβέρνηση. Βεβαίω η δική σας επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως και σε πιθανές μεταρρυθμίσεις ε, της συνθήκης ε, της Λισαβόνας και γι' αυτό θα πω και δύο λόγια και ε, για αυτό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως με τον Αντώνιο Βιτορίνο όταν ε, λέει ή μάλλον ε, αντίθετα με αυτόν, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονα σε θεσμικά ζητήματα ε, θα γνωρίζετε ίσως ότι ο Αντώνιο Βιτορίνο μαζί με τον Μισελ Μπαρνιέ εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Συνταγματική Συνέλευση. Επομένως, ε, ε, ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάει όταν αναφέρεται στα θέματα αυτά. Κάτι το οποίο και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μας αναφέρει αυτά τα θέματα. Και συμφωνώ απολύτως ως προς το γεγονός ότι προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση Πλήρω των δυνατοτήτων τη εθήκης της Λισαβόνας για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητο να αποκαταστήσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Βορρά και Νότου της Ευρώπης, ε, Δύσης και Ανατολής επίσης. Και ε, θεωρώ ότι το θεσμικό όργανο το οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω για 10 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιδίω αυτή τη στιγμή που θέλει να αποκαλείται και άλλοι θέλουν να το αποκαλούν μια πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να κάνει τα ουσιώδη του πολιτικού έργου, που κατά την άποψή μου δεν είναι να εκπέμπει δόσεις ευελιξίας βάσει των ισορροπιών δυνάμεων, αλλά να αποτανθεί στους ηγέτες των κρατών μελών με πολιτικό τρόπο, χωρίς ε, ε, καμία διανοητική πολιτική υποταγή και να κάνει προσπάθεια προκειμένου να πείσει τους ηγέτες των κρατών μελών ότι αυτό το οποίο τους διαιρεί ναι μεν υπάρχει, αλλά ε, τίνουν ο καθένας από αυτούς ε, να το βλέπει στην υπερβολή του. Και ε, το λέω αυτό διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό το ε, παιχνίδι των προκαταλήψεων. αν δούμε τους τρεις βασικούς πυλώνες κατά την άποψή μου της οικονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο απαιτείται είναι μια κοινή δέσμευση ώστε ε, να υποστηρίξουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο, κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να το αναδιαρθρώσουμε, αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε ουσιαστικά. Και μέσω ουσιαστικής βελτίωσης εννοώ κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ πιο σημαντικό από τις ε, βελτιώσεις ε, που είναι πολύ σημαντικές ε, που προτείνει η επιστολή των πέντε προέδρων. Η βασική βελτίωση είναι να δούμε ποια είναι τα εκρεμή εμπόδια για την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη, που είναι πιο θεμελιώδη όμως, διότι εδράζουν στις ε, τεράστιες αποκλήσει που υπάρχουν μεταξύ των διαφέρων πολιτικών νοοτροπιών. Ε, εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση ως εξή. Υπάρχουν τρεις βασικές τάσεις. Η μία τάση είναι μεταξύ ολοκλήρωσης της αγοράς ε, και ε, κοινωνικών συνεπειών, εθνικών συνεπειών ε, και όλα αυτά κατά της ολοκλήρωσης. Αυτές οι εντάσεις καθυστερούν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και έτσι οδηγούν σε λιγότερη ολοκλήρωση και σε μικρότερη ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει μεταξύ δημοσιονομικών κανόνων και ευελιξίας. Αυτή η ένταση δημιουργεί αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης σε δύο διαχωριστικές γραμμές και γεωγραφικά μέσω βορρά και νότου αλλά και πολιτιστικά μέσω του ε, γερμανικού ορθοφιλελεύθερου οράματος και του αγγλοσαξονικού οράματος. Οι εντάσεις αυτές αφενός αυξήνουν τι εντάσεις για την εφαρμογή του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη και ε, αφετέρου δημιουργούν προβλήματα σε εθνικό επίπεδο ε, και δεν επιτρέπουν να υπάρχει ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο που κανονικά θα έπρεπε να, έρχεται, να βοηθήσει τις επενδύσεις για την εφαρμογή του σχεδίου Juncker. Και η τρίτη ε, τάση την οποία μελετώ πρόσφατα είναι η τάση και η ένταση μεταξύ αυτών που είναι ε, καθαροί δικαιούχοι και αυτών που είναι καθαροί χορηγοί. Αυτή η ένταση, η οποία δηλητηριάζει τη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως έχει, ο προπολογισμό είναι μάλλον παροχημένος ε, για τις διαρθρωτικές δαπάνες, δεν είναι διάφανος, δεν είναι δημοκρατικός και είναι ε, οπισθοδρομικός στον τρόπο χρηματοδότησης. Αυτό λοιπόν το οποίο ονειρεύομαι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερμηνεύοντας τη φύση της ως πολιτική επιτροπή με την πιο ε, ευγενή έννοια που νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο με το πολιτικοποιημένη είναι να έχει τέτοια σχέση με τις, τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν να βρουν ποιο είναι ο κοινό τόπος που έχουν που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα κοινή δέσμευση για την ε, ε, ολοκλήρωση και την ανάπτυξη να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία ε, θεωρώ ότι κατά την άποψή μου απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν κάποια πράγματα και δεν είναι αδύνατα. Ε, για 1,5 χρόνο ε, ήμουνα μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύντομο διάστημα, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εάν τρεις ή τέσσερις ηγέτες από ουσιαστικές βασικές χώρες της Ευρωζώνης καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για μισή μέρα, μια μέρα. Θα καταλήξουν σε μια θέση που θα μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ τους. Όχι μόνο γιατί θα έχουν ένα κομψό τελικό ανακοινωθέν, αλλά γιατί πραγματικά θα υπάρχει μια βαθύτερη, πραγματική ε, αντίληψη των κοινών θέσεων. Και αυτή η συζήτηση είναι αυτή η οποία επέτρεψε στις πολιτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη Σύνοδο του Ιουνίου του 2012 να συμφωνήσουν ομόφωνα, κυρίως ε, στη Σύνοδο της Ευρωζώνης, Γεγονός που επέτρεψε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να πει μερικές εβδομάδες αργότερα αυτά τα οποία δήλωσε, δηλαδή ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπεριέλαβε αυτή τη δήλωση ουσιαστικά στην απόφαση για το νέο ε, αυτό μέσο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει για κάθε μία από αυτές τις τρεις διαφορετικές εντάσεις ε, να μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο. Για την ενιαία αγορά, την πρώτη ένταση που υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα συμφιλίωση μεταξύ της αγοράς και των κοινωνικών συνιστοσών της οικονομίας της κοινωνικής αγοράς. Βλέπω να μπαίνει ο κύριος Μπροκ, επομένως η οικονομία της κοινωνικής αγοράς ε, μου ήρθε αυθόρμητα ως όρος εντελώς αυθόρμητα μόλις σας είδα κύριε Μπρόκ. Η αγορά και οι κοινωνικές συνιστώσεις της ε, κοινωνικής ε, ε, αγοράς θα πρέπει λοιπόν να συμφιλειωθούν πολύ περισσότερο και για να μπορέσουμε να άρουμε κάποια από τα προσκόμματα τα οποία θα βοηθήσουν την ταχύτερη έγκριση της νομοθεσίας για την ενή αγορά και κατά συνέπεια και την εφαρμογή της, πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος μεταξύ άλλων για ε, μια ήπια αλλά αποτελεσματική πολιτική συντονισμού σε φορολογικά θέματα. Και αυτή η πολιτική θα πρέπει ε, να γίνει κάπως λιγότερη δύσκολη και μάλλον αυτό θα το καταφέρουμε όταν τα βασικά κράτη-μέλη τα οποία παραδοσιακά αντιτίθενται περισσότερο από άλλα ε, δεν θα είναι πλέον στο τραπέζι της λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ε, όταν διατυπώθηκε, κατά πάσα πιθανότητα ήταν το κατάλληλο τότε δηλαδή που ξεκίνησε το ευρώ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευτυχή θέση, εάν αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα ως έχει, να έχουμε την αξιοπιστία του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο μηδέν. Απατώμαστε ικτρά όταν συζητούμε για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εγώ είμαι Ευρωπαίος, ε, Νότιο Ευρωπαίος, ο οποίος δεν θα ήταν ικανοποιημένος εάν οι αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας ε, ε, διαγράφονταν παντελώς. Αυτό θα ήταν εθνική χαρά για κάποιες χώρες, αλλά και εθνική καταστροφή μακροπρόθεσμα στις ίδιες αυτές χώρες. Αυτή τη στιγμή όμως η παρούσα κατάσταση είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει σοβαρή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και αυτή λοιπόν είναι η ιδανική στιγμή να μπορέσουμε να βάλουμε γύρω από ένα τραπέζι το βορρά και το νότο και να παραδεχτούμε ότι αφενός όλες αυτές οι δόσεις ευελιξίας ε, που τις περισσότερες ε, περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για τις τρέχουσες δαπάνες σε εθνικό επίπεδο ε, δεν θα πρέπει να υφίστανται, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει όλοι να δούμε με πιο ευνοϊκό μάτι και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό τι εθνικέ δημόσιε επενδύσει. Με τη στενή του έρια ε, ε, ε, έννοια να εφαρμόζονται αυστηρά ώστε να μην υπάρχουν εντερτύπια. Αλλά δεν μπορούμε να ελπίζουμε να επανεκκινήσουμε σοβαρά την ευρωπαϊκή οικονομία εάν έχουμε μόνο το σχέδιο Juncker το οποίο καλώς καμωμένο, αλλά ε, δεν υπάρχει και κάτι ε, το οποίο θα βοηθήσει τις δημόσιες επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο. Ακόμα και με γερμανικές αρχές δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε ότι Εάν ε, δεν μπορούμε να δανειστούμε λίγο περισσότερο από τις αγορές όταν στοιχίζει 0%-0,5% ώστε να έχουμε μια καλύτερη πρικοδότηση υλικών και άειλων υποδομών για τις μελλοντικές γενιές των Γερμανών και των Ευρωπαίων, είναι μια λογική πρόταση. και ουσιαστικά κινούμαστε κατά των νέων γενεών εάν δεν το κάνουμε αυτό. Και τέλος, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, νομίζω ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να επικεντρωθούμε και πάλι, ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί και πάλι στα ουσιώδη, αυτά που κάνει καλά. Και τώρα το βασικό αίτημα είναι να δοθούν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, να υπάρχει έλεγχος αλλά και συνδρομή προς τους μετανάστες. Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που τα κράτη-μέλη στρέφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λένε ότι θα πρέπει να το κάνετε εσείς αυτό γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως η άποψή μας ε, στην ομάδα υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους που θα ε, παρουσιάσει και την έκθεσή της εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα δύο άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Ιανουαρίου, θα είναι ότι εάν τα κράτη-μέλη συμφωνήσουν ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν νέες ίδιες λειτουργίες, δεν θα ήταν και εξωπραγματικό να πιστέψουμε ότι όντως υπάρχουν και νέοι ίδιοι πόροι για αυτές τις νέες ίδιες, ε, ε, τα νέα ίδια καθήκοντα, ε, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Μια τελευταία παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω κάποια πρόταση να σας κάνω όσον αφορά μια πιθανή νέα συνθήκη. Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι εάν δεν γίνει αυτή η προσπάθεια, οι διάφορες πολιτικές νοοτροπίες να προσεγγιστούν, θα ήταν άχρηστη ακόμα και η συνθήκη. Και αν γίνει αυτή η προσπάθεια με επιτυχία, μπορεί να μην χρειάζεται νέα συνθήκη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προτείνω και το πιστεύω ακράδαντα είναι ότι όλη η θεσμική εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο αλλά και η Ευρώπη εν γέννη θα πρέπει να εστιάσει σε μία ίσονη σημασία πτυχή πριν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση για νέα συνθήκη. Γνωρίζουμε όλοι εδώ και χρόνια ότι η διαδικασία κύρωσης όσο έχει αυτή τη στιγμή είναι μοιραία επιβάρυνση για οποιαδήποτε αναθεώρηση της συνθήκης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός ο θεσμός της αμεσοδημοκρατίας, ε, το δημοψήφισμα, έδειξε το δύσκολο πρόσωπό του στη Δανία, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, ε, στην Ολλανδία και στην ενσάρκωσή του κάθε φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια άλλε εμπειρίε δεν έχουν δείξει καλύτερη ή μεγαλύτερη ευκολία και απλότητα και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στο δημοψήφισμα για το Brexit. Αλλά χρειάζεται στα αλήθεια ακύρωση μέσω αυτής της διαδικασίας. Θυμάμαι μια περίπτωση για την δική μας την Ευρώπη, τον Νότερ Ρόπ, που τότε προείδρευε ο Τομάζο Πάμπλιας και όταν με τον οποίο συζήτησα τα θέματα αυτά. Και εγώ, διότι εγώ έγραψα αυτό το άρθρο, ε, παρουσιάσαμε μια διαφορετική μέθοδο. Εγώ δεν είμαι νομικός βέβαια, πιστεύω ότι οι νομικοί θα πρέπει να διερευνήσουν κατά πόσο ε, είναι παντελώ αδύνατο να έχουμε μια διαφορετική διαδικασία κύρωσης. Η ιστορία είναι με το μέρον μας, διότι μας λέει ότι δύο χώρες στις δύο πιο γνωστές ομοσπονδίε στον κόσμο δεν κύρωσαν το σύνταγμα το οποίο ισχύει για τις ομοσπονδίες τους. Το Ροντ Island η πολιτεία του Ροντ Island και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε. Η πολιτεία του Ροντ Island λοιπόν που δεν συμμετείχε στις συζητήσεις ε, της ε, ε, συνθήκης της Φιλανδέλφειας και απέριψε το κείμενο την πρώτη περίπτωση που ήρθε να προσθεθεί ε, στην άλλη πολιτεία των, ε, μάλλον, στις υπόλοιπες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που έλυσαν να την αποκλείσουν. Και στη Γερμανία ε, το ελεύθερο κρατήδιο της Βαβαρίας το 1949 αρνήθηκε την κύρωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αλλά με ένα ρεαλισμό τον οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε δέχτηκε ε, την εφαρμογή του στη βαβαρική επικράτεια. Και αυτό είναι παιχνίδι γιγάντων ε, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τη Βαβαρία. Ένα ενδεχόμενο που είχα ε, προτείνει σε εκείνο το έγγραφο πριν από 10 χρόνια ήταν το εξής. Όταν υπάρχει μια νέα συνθήκη, η οποία υπογράφεται εξ ορισμού από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κάθε κράτους μέλους, θα πρέπει επίσης να υπάρχει και ένα επιπλέον άρθρο, το οποίο θα υπογράψω καθής εξ αυτών, και θα λέει ότι στην περίπτωση που στη χώρα μου αυτή η συνθήκη, την οποία έχω υπογράψει εγώ, δεν περάσει από τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής κύρωσης ή από τη διαδικασία του δημοψηφίσματος και δεν γίνει αποδεκτή, εγώ σας διαβεβαιώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι σε έξι μήνες από εκείνη την ημερομηνία θα υποβάλω προς κύρωση μία δεύτερη πρόταση, η οποία θα λέει, ή μάλλον θα θέτει το ερώτημα στους πολίτες, θέλετε η χώρα μας να παραμείνει ε, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το συνταγματικό αυτό κείμενο το οποίο έχουν κυρώσει σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι ή προτιμάτε να αποχωρήσουμε. Αυτό μπορεί να φέρει και τους πολίτες αντιμέτωπους με μια ριζοσπαστική εναλλακτική λύση. Είχαμε μια πρόσφατη εμπειρία ριζοσπαστικών εναλλακτικών λύσεων αλλά αυτό το οποίο προτείνω είναι ότι, μάλλον λέω, ότι ε, τα μεγαλύτερα μυαλά της πολιτικής Ευρώπης θα πρέπει ε, να μην κάθονται να σκέφτονται τόσο στο 100% τι θα περιλαμβάνει μια νέα συνθήκη, διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει από όλα τα φίλτρα της διαδικασίας κύρωσης, αλλά κατά πόσον υπάρχουν ε, νομικές και πολιτικά πιθανές λύσεις να ε, εγκριθούν άλλα πράγματα, άλλοι τρόποι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοντή. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να σχολιάσουν και τις απόψεις του κυρίου Μόντι, υπέρ των οποίων εκφράζεται και η έκθεση, καθώς επίσης και το, ε, υπόλοιπες απόψεις που ακούσαμε. Κύριε Μερσέντες, πρέσα, θα μιλήσω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τους ε, δύο εισηγητές για την ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μόλις ξεκίνησε. Σε πολλούς από εσά έχουμε ήδη υποβάλει την έκθεση ε, στο αρχικό της στάδιο, θα το θυμάστε άλλωστε. Εγώ λοιπόν εδώ θα περιοριστώ να σας πω κάποιες σκέψεις και να σας πω και δύο λόγια για την εξέλιξη της ε, έκθεσης. Καταρχάς, όπως ε, ε, υπενθυμίσαμε, εμείς γνωρίζουμε ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Καταρχάς, να αποκτήσει και πάλι μια πιο δημοκρατική ε, θεσμική δομή που θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις ε, απαιτήσει των πολιτών, αλλά να ανταποκριθεί και ταχύτατα στις προκλήσεις του εξωτερικού κόσμου, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Είναι σαφές ότι υπάρχουν συνεπώς μια σειρά από πτυχές οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν. Καταρχάς, η δημοκρατικότητα της διαδικασίας, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς, αλλά και οι νέες προκλήσεις, ιδίως εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τις εξωτερικές δράσεις, με την άμυνα, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Είναι οι πιο πρόσφατες ε, προκλήσεις, ε, εξίσου σημαντικές όμως, και όλες μπορούμε να τις εντοπίσουμε σε μεγάλο βαθμό με τα μέσα τα οποία μας διαθέτει η συνθήκη. Ένα πρώτο τμήμα της έκθεσής μας αφορά τις πιο θεσμικές πτυχές. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η κοινοτική μέθοδος είναι μακράν καλύτερη της διακυβερνητικής μεθόδου, διότι η διακυβερνητική μέθοδος είναι ένας από τους λόγους όχι μόνο για τις καθυστερήσεις, αλλά και για τις απαιτυχίες και τις δυσκολίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ε, αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερο. Επομένως, ε, υπενθυμίζουμε ότι η συνθήκη προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες μέσω της ε, ρήτρας Πασερέλ αλλά και μέσω άλλων εργαλείων. Δεν ε, υπάρχει λόγος να εμβαθύνω πολύ, αλλά εμείς ε, θεωρούμε ότι από αυτήν την άποψη υπάρχουν μια σειρά από πτυχές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε. Η πρώτη αφορά κυρίως ε, τη λειτουργία του Συμβουλίου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως όμως του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει μέσα βάσει της συνθήκης ε, να μοιάζει όλο και περισσότερο με μια ευρωπαϊκή γερουσία. Πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως μπορεί άλλωστε να το κάνει, αλλά να το κάνει σπανίως, ε, την ε, ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Και επίσης ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει αφενός να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και η μεγαλύτερη αυτή η διαφάνεια ε, μπορεί να προκύψει αν υπάρχει μόνο μία νομοθετική σύνθεση και όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις να είναι κάτι αντίστοιχο με τις μόνιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι θα ήταν πιο ε, σαφής ο άλλος πυλώνας του δημοκρατικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτι που είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των πολιτών που πιστεύουν ότι τα αποφασίζει όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε πότε διαδραματίζει κάποιο μικρό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο είναι κρυμμένο σε ένα νέφος πλήρους άγνοιας. Επομένως, η διαφάνεια του Συμβουλίου στην ομοθετική του δράση θεωρούμε ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Η δεύτερη πτυχή που αφορά πρωτίστως ε, τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίως ε, μια μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου, επαλήθευσης της δράσης των κυβερνήσεών τους όταν συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία ή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στι συμβαστικέ ε, τροπολογίε, είναι σχεδόν έτοιμε οι συμβαστικέ τροπολογίε γιατί θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα τα οποία ακριβώς προσπαθούν να αντιληφθούν λίγο καλύτερα πώς θα μπορούσε να ε, λειτουργήσει η κοινή εργασία μετά την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 13 όπως την αποκαλήσαμε για να είναι πιο δημοκρατική η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές οικονομικής πολιτικής, οι οποίες δεν θα είναι αυστηρά ε, δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, ε, πολιτικής εργασίας, ώστε ο έλεγχο από πλευρά εθνικών κοινοβουλίων για τις πολιτικές των κυβερνήσεών τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη μια να είναι ευρύτερο και ε, να καθορίζεται σαφέστερα βέσω μία συζήτησης ε, για τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, ε, για τις διάφορες οικονομικές πολιτικές. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που αφορούν το ρόλο των κοινοβουλίων, αλλά όλο αυτό το θέμα είναι τμήμα μιας δέσμης προβληματισμών για το πώς μπορούμε να έχουμε μια στενότερη σχέση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική ευθύνη αλλά και η δημοκρατική προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε και τη δυνατότητά μας να απαντούμε από κοινού στις απαιτήσεις των πολιτών μας. Υπάρχει όλο αυτό το σκέλος το οποίο αφορά την οικονομική πολιτική. Οι συνάδελφοι επικεντρώθηκαν πολύ στο θέμα αυτό και και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι είναι απόλυτα σωστό το θέμα της σύγκλησης των οικονομιών αλλά και της ευθύνης των κυβερνήσεων. Πιστεύουμε όμως ότι το πέρασμα από έναν απλό συντονισμό πολιτικών, δημοσιονομικών πολιτικών με κάπως αυστηρές προδιαγραφές και να φτάσουμε σε ένα πραγματικό κώδικα σύγκλησης που θα περιλαμβάνει και μία σειρά από στοιχεία τα οποία δεν είναι αμυγός ε, οικονομικά και ε, ε, χρηματοπιστωτικά, αλλά να υπάρχουν και κάποια πράγματα που αναφορούν εργασιακά ζητήματα. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα μας επιτρέπει να πούμε στους πολίτες ότι δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε πτυχές οικονομίας που αφορούν την εσωτερική αγορά, αλλά είναι μια σύγκληση που αφορά ευρύτερα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, δεν έχω χρόνο, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πορεία επιτρέπει να έχουμε και πολιτικές πειθαρχίες οι οποίες είναι μεν απαραίτητες αλλά να τις κατανοούν και να τις αποδέχονται αυτές οι πολιτικές οι πολίτες γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να τις επιβάλλουμε. Υπάρχει και ένα τμήμα ε, αρκετά μακροσκελές και πολύ σημαντικό το οποίο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά όσον αφορά τη δυνατότητα βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέσα τα οποία υπενθυμίσαμε πρόσφατα. Για παράδειγμα τα, τα ανέφερε η καγκελάριος Μέρκελ, οι Υπουργοί Άμυνα, οι οποίοι ε, συναντήθηκαν στην Πρατισλάβα. Υπάρχουν μέσα λοιπόν εντός της συνθήκης που μας επιτρέπουν να κινηθούμε προς μια πολιτική ε, ε, σε εξωτερική πολιτική και πολιτική κοινή ασφαλείας, ε, κυρίω όσον αφορά την άμυνα, η διαρθρωμένη συνεργασία, η ενισχυμένη συνεργασία, η οποία είναι γνωστή. Η συνθήκη περιλαμβάνει πληθώρα ευκαιριών και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι μας πιέζουν τόσο πολύ τα χρονικά περιθώρια που η χρήση της συνθήκης της Λισαβόνα στον τομέα αυτό ου μόνον είναι πιθανή, αλλά ε, είναι ολοένα και πιο απαραίτητη. Επομένως, ακόμα και οι πολιτικές ε, για την αντιμετώπιση την, ε, της τρομοκρατίας και πολιτικές πέτσες ασφάλειας, ε, όπως επίσης και η βελτίωση της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, είναι δυνατές βάσει της συνθήκης και θεωρούμε ότι αποτελούν μία πρόκληση την οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποδεχθούμε. η συνθήκη, όπως ξέρετε, ήταν μια συνταγματική συνθήκη που περιλέμβανε ένα ε, αμάλγαμα δυνατοτήτων που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια. Διότι ε, η όθηση για να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν θα είναι η συγκέντρωση πολλών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να ξεκαθαρίσουμε τις βασικές αρμοδιότητες που θέλουμε να διαχειριστούμε από κοινού και να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε από κοινού να ανταποκριθούμε τα όσα μας ζητούν οι πολίτες μας με δημοκρατικό τρόπο. Να γίνει δηλαδή πιο δημοκρατική αυτή η διαδικασία θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο στοιχείο ε, που περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας μέσω των διαφόρων μέσων που και σε αυτή την περίπτωση δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς. Ε, θα σταματήσω εδώ. Ε, αυτά είναι τα γενικά θέματα. Αν θέλετε να συζητήσουμε λεπτομέρειες μπορούμε κάλλιστα να τις συζητήσουμε. Θα ήθελα απλό ε, να, πω ότι για τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, εμβαθύναμε πάρα πολύ αυτές τις πτυχές, εξετάσαμε πιο διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα άρθρα της συνθήκης μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και επίγουν. Ευχαριστώ πολύ. So, uh, you... Σας ευχαριστώ. Έλμαρ, που προσθέλετε το λόγο. Και μετά θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάποια πράγματα. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω με το παράδειγμα που είπε ο Μάριο Μόντι που μίλησε για την ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς. Θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην εξέβρεση ισορροπιών στον οικονομικό τομέα και τον κοινωνικό τομέα. Και θα τις βρούμε μόνο εάν διαμορφώνουμε σωστή πολιτική. Ε, και εάν ε, εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, αν δεν έχουμε σωστή επιβολή του νόμου, δεν ε, θα το πετύχουμε αυτό. και μπορεί το μισό του κοινοβουλίου να λέει ένα πράγμα και το άλλο μισό να λέει άλλο. Χρειαζόμαστε όμως να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή σχέση ανάμεσα στην νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικές μεθόδους λήψης αποφάσεων. Εάν συμφωνήσουμε ως προς αυτές ε, τις πιο ε, αποτελεσματικές μεθόδους, ε, πώς θα πετύχουμε και την νομιμοποίηση. και την αποδοχή από το κοινό. Νομίζω ότι δύο πράγματα απαιτούνται εδώ. Καταρχάς, θα πρέπει να καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντα και να πούμε ποια από αυτά μπορεί να λύσει καλύτερα η Ευρώπη και πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της επικουρικότητας υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που δεν μπορούν να λύσουν μόνα τους ε, τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε έλλειψη ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, αδιαφορία για την Ευρώπη ε, και αντίθεση προς την Ευρώπη. Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο και δεν μπορούμε να βρούμε την έξοδο. Γι' αυτό θα ήθελα να πω το εξής που μας απασχολεί τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες. Ε, έχει να κάνει με την επικύρωση της συμφωνίας ΣΥΤΑ. Το θέμα δεν είναι αν βρίσκουμε σωστή ή λάθος τη συμφωνία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για κάτι, τότε θα πρέπει να θεωρείται ότι η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει και την απαραίτητη νομιμοποίηση. Εάν διαχωρίσουμε το επίπεδο ε, λήψης αποφάσεων από το επίπεδο νομιμοποίησης, ε, τότε έχουμε πρόβλημα. Και θέλω να είμαι σαφής. Ε, υπήρχαν εσωτερικές αντιθέσεις, είχαμε εθνικές διαμαρτυρίες και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια στη δικασία λήψης αποφάσεων, αλλά ε, έτσι τελειώνει όλη η υπόθεση. Εάν έχουν δοθεί αρμοδιότητες ε, στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει και ένα άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα Συμβούλιο το οποίο ε, έχει την ομοποίηση από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, θα πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτές. Και αν δεν γίνονται δεκτές αυτές οι αποφάσεις θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα τότε θα πρέπει νωρίτερα να έχουμε συζητήσει εάν θέλουμε να, να εκχωρήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες στην Ευρώπη. Ε, αλλιώς σας πει το εθνικό επίπεδο ότι εμείς μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να αφήσουμε απ' έξω την Ευρώπη. Όχι όμως να έχουμε ένα τέτοιο μείγμα. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες ε, και γι' αυτό προτείνουμε εγώ και η κυρία Μπρέσο ε, μεταρρύθμιση στο Συμβούλιο. Είδαμε το Brexit επειδή επί 10 χρόνια εξηγούν στους πολίτες ότι η Ευρώπη είναι κακό πράγμα δεν θα πρέπει ε, τώρα να μας εκπλήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Και γενικά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά φταίει η Ευρώπη, ενώ όταν ε, πάνε καλά τα πράγματα, ε, τότε ε, αυτό είναι, αυτό οφείλεται στα εθνικά κοινοβούλια. θα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πιστεύουμε ότι με απλές τροποποίησεις του κανονισμού του Συμβουλίου μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Στο, ε, στη συνθήκη λέει ε, το ε, Συμβούλιο Υπουργών, όχι τα Συμβούλια Υπουργών. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως δεύτερο νομοθετικό σώμα θα πρέπει να συνεδριάζει ανοιχτά και να ενημερώνει τους πολίτες ε, σχετικά με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, ώστε όλα να είναι διαφανή. Έτσι, τα επιμέρους σε Συμβούλια Υπουργών μπορούν να είναι οι επιτροπές που θα συζητάνε εσωτερικά. Αλλά αυτή η διαφυγή των εθνικών, κοινοβουλίων, ε, των εθνικών κυβερνήσεων από ε, την ευθύνη τους ε, νομίζω ότι είναι ένα ε, θέμα που θα πρέπει να λύσουμε. Αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Μερσέντες αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Όταν έχουμε κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, θα πρέπει αυτές ε, να έχουν και δημοκρατική νομιμοποίηση και αυτή η νομιμοποίηση θα πρέπει να διασφαλίζεται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ισχύουν για 4 ή 6 χρόνια οι κατευθυντήρες γραμμές αυτές. Θα πρέπει Ε, στην ε, Ευρώπη ε, όταν έχουμε την διαδικασία με έλεγχο κλπ. να αναλαμβάνουν και τα εθνικά κοινοβούλια τις ευθύνες τους. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια, το καθένα όμως στο επίπεδό του. Ε, δεν θέλουμε να έχουμε αδιαφανείς καταστάσεις και έλλειψη αποτελεσματικότητας. Ε, βλέπουμε ότι όπου συζητάμε εθνικό χρήμα, αποφασίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, έχουμε εθνική αρμοδιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό. έχουμε εξαμηνιαία διάσκεψη μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα αμήνης που λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ο καθένας γνωρίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του και έχουμε ένα καλό σύστημα επικοινωνίας. Και έχουμε και τρόπο να ελέγχουμε και τις διάφορες αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο αμοιβαίος έλεγχος και η λογοδοσία. Πιστεύω ότι αυτή η διάσκεψη με βάση το άρθρο 13 αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με καλύτερο τρόπο. Ε, και ε, ευχαριστώ για όσα υπόθηκαν σχετικά με τις δυνατότητες μεταρρύθμισης. Ε, πράγματι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν την παγίδα. Η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ε, δεν δεσμευόμαστε από την ομοφωνία. Γνωρίζουμε ότι ισχύει αυτή τη στιγμή η ομοφωνία και ότι μάλλον είναι <coughs> δύσκολο να την παρακάμψουμε. Ξέρουμε ότι το σταματικό Δικαστήριο της ε, Γερμανίας έχει λάβει προβληματική απόφαση όσον αφορά την απόφαση ΣΥΤΑ και αυτό είναι πιο προβληματικό από την στάση της Βαλονίας. Θα πρέπει όμως να διαπιστώσουμε ότι η ομοφωνία αποτελεί πρόβλημα και η Βαβαρία ε, ακόμα και σήμερα δεν έχει ε, επικυρώσει την ε, συνθήκη διότι ε, επικαλείται την αρχή της επικουρικότητας. Πώς όμως ε, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα να μην θίγεται η κυριαρχία των κρατών μελών, ε, από την άλλη όμως ε, να υπάρχει η δυνατότητα δράσης. Ο συνάδελφος ε, Βιτορίνη θα θυμάται την συνταγματική συνέλευση. Εκεί θέλαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα, αλλά δεν το καταφέραμε. Η έκθεση Φερχόφστατ προτείνει να ξαναεξετάσουμε το θέμα. Υπάρχει όμως και η έκθεση η δική μου μαζί με την κυρία Πρέσο, Πρέσο Πρόκ, ε, που ασχολείται με την ρήτρα γέφυρας, ε, το Passerelle Clause. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, η Ευρώπη μπορεί να λύνει από κοινού προβλήματα χωρίς να μπλοκάρεται από έναν μόνο. Η συνθήκη με την διευρυμένη συνεργασία προβλέπει εργαλεία ώστε να μπορεί να προχωρεί μία ε, συνεργασία των προθήμων. Αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει θα πρέπει να, επιτρέψει θα ήταν δίκαιο να ε, επιτρέψει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο και να μην ε, χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αρνησικήριας του. Αυτή λοιπόν η συνεργασία των προθήμων θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μην δημιουργηθούν πρόσθετα εμπόδια. Το ίδιο ισχύει για το Σέγγεν, για το ευρώ επίσης ε, και ο Ζακ Τελόρ είχε αναφερθεί σε αυτό. Το να δημιουργούμε νέους φορείς εντός ε, της Ευρώπης ε, δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία και επίσης δημιουργεί διαιρέσεις. Δεν ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες δομές. Θα πρέπει να βρούμε πιο ανοιχτούς δρόμους. που να σέβονται την βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε την ισότητα για να λειτουργήσει καλά. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε εδώ μια κατάλληλη προσέγγιση. Ο Μάριο Μόντι, με ευκαιρία το δημοψήφισμα, είπε ότι μέσα στα δύο τελευταία χρόνια ε, ε, έχω γίνει ε, πολύ αντίθετος με τα δημοψηφίσματα και Ε, είδα στη χώρα μου την αποτυχία της δημοκρατίας μετά τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Και αυτό έγινε με δημοψηφίσματα ε, τέλη της δεκαετίας του 20, αρχές δεκαετίας του 30. Ε, εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν οι αρχές τα δημοψηφίσματα για να διαλύσουν τις δημοκρατικές δομές. Και όταν βλέπω ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν στα δημοψηφίσματα, Βλέπουμε στην Ιταλία το θέμα που φαίνεται να καταλήγει στο αν ε, αρέσει σε κάποιον ο Ρέντσι ή όχι. Χρησιμοποιούνται λοιπόν τα δημοψηφίσματα για να υπονομεύσουν ε, την δημοκρατία και αποτελεί τρόπος να διαφύγουν ε, οι πολιτικοί από τις δικές τους ευθύνες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη οδός να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Εννέα συνάδελφοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών και μπορώ να σας δώσω εύκολα μέχρι και πέντε λεπτά. Βεβαίως αν δεν ακρηγορήσετε ακόμα καλύτερα αλλά ε, σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις σας για αυτά που εξέφρασαν οι τέσσερις ε, ομιλητές μέχρι τώρα. Βεβαίω, αν λάβω και άλλες, ε, άλλα αιτήματα εγγραφή στον κατάλογο των ομιλητών, θα χρειαστεί να αλλάξω και το χρόνο ομιλίας. Επομένως, προσπαθήστε να το υποβάλλετε αυτά τα αιτήματα τώρα. Ας ξεκινήσουμε με τον με τον κύριο Στάουτ από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίση. Συμφωνούμε ως προς αυτό. Θα πρέπει όμως επίσης να εξετάσουμε ποιες είναι οι αιτίες για την κρίση αυτή, τι μας έφερε στην κατάσταση αυτή. Βλέπουμε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ε, αντιδρούν πια όπως περιμένουν οι πολίτες ότι θα αντιδράσουν. Και το χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Και αυτός είναι ο λόγος ε, που οι πολίτες πιστεύουν ότι όσα συμβαίνουν δεν είναι προς συμφέρον τους. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε είναι ποιος ευθύνεται για την εξέλιξη αυτή. εάν απαντήσει κανείς ότι οι πολίτες φταίνε ότι εκείνοι είναι υπεύθυνοι, αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Οι πολιτικοί θα πρέπει να εκπροσωπούν ε, τους πολίτες ε, αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η δημοκρατία διαλύεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κοινοβούλια μπορούν να προσπαθήσουν να έρθουν περισσότερο σε επαφή με τους ανθρώπους και να τους δείξουν ότι όσα συμβαίνουν, συμβαίνουν προς συμφέρον τους. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες πιστεύουν ότι χρειάζεται ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αρκετοί ομιλητές. Ήδη ανέφεραν κάποιες πιθανές λύσεις. Η κίτρινη κάρτα μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Στην πράξη όμως δεν λειτουργεί. Με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, 11 χώρες, 11 κοινοβούλια δεν ε, έχουν ε, συμφωνήσει και χρειαζόμαστε πιθανότατα νέα συνθήκη, αλλά αυτή τη στιγμή εντός της ε, ισχύουσας συνθήκης δεν δίδεται η νομική βάση για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Η Κομισιόν θα πρέπει να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας των συνθήκων. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης, διαπιστώσαμε ότι επέκριναν διάφοροι την ε, Ουγγαρία επειδή προσπάθησε να προστατεύσει τα σύνορά της. Και μάλιστα μας κατηγόρησαν κράτη τα οποία τα ίδια έχουν ε, παραβιάσει ε, κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, έχουμε το θέμα των λόμπι, των ομάδων συμφερόντων. Ε, αναφέρεται συχνά ότι η Ευρώπη είναι θύμα των ε, λόπις, ε, τίποτα δεν είναι ρυθμισμένο. Συζητήθηκε και πολύ ο πρόεδρος της Επιτροπής που μετά το τέλος της θητείας του εργάζεται σε μεγάλη πολυεθνική. Ε, να σας δώσω ε, ως παράδειγμα την Ελβετία. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η Ελβετία δεν είναι δημοκρατική χώρα. Η χώρα όμως ε, είναι έτσι δομημένη που σε ομοσπονδιακό επίπεδο λύνονται θέματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν μόνα τους ε, τα καντόνια. Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς λειτουργεί η Ελβετία. Ίσως θα μπορούσαμε να μάθουμε από το παράδειγμά της. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Δώδεκα τελικά θα είναι οι ομιλητέ, επομένω θα ήθελα να σα ζητήσω να περιοριστείτε σε 4 λεπτά ομιλία ο καθένα. Ο κύριος ε, Βαν Χόλικ ε, από την Ουγγαρία επίσης. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω ότι υπάρχει κοινή κατανόηση ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου είναι απολύτως απαραίτητο να εξετάσουμε, να επανεξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επικροτούμε τη διαδικασία που ξεκίνησε στην Μπρατισλάβα, διότι νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο ανοιχτά και ειλικρινά να εξετάσουμε που υπάρχουν ε, ε, αντιθέσεις, αποτυχίες κλπ. Ο κύριος Βιτορίνο είπε ότι πιθανότατα είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη δεν βγαίνει ε, ενδυναμωμένη από μία κρίση και ότι μπορεί να διαλυθεί. Πώς λοιπόν μπορούμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί ε, να γίνει αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Η δική μας ε, θέση είναι ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην Ευρώπη. Ε, δεν θέλουμε όμως να εθελοτυφλούμε, να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Θα πρέπει να βρούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να κολλήσουμε σε ιδεολογίες, θα πρέπει να βρούμε λύσεις στα προβλήματα. Το κείμενο της ε, Mercedes Presso και του Elmar Brock ε, περιέχει πολύ καλές ε, προτάσεις και ρεαλιστική προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι Σήμερα εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ε, δύο διαφορετικές απόψεις όσον αφορά ε, τον τρόπο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε την ε, ομοσπονδιακή προσέγγιση και έχουμε την ευρωσκεπτικιστική προσέγγιση. Βλέπουμε κάποια παλιά αντανακλαστικά. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πολλοί λένε ότι χρειαζόμαστε εμβάθυνση της Ένωσης, χρειαζόμαστε ε, πιο βαθιά Ένωση. Υπάρχει όμως ε, και μία τρίτη αντίδραση, να εξετάσουμε τα ε, προβλήματα με πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο και να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι αν ε, αποτύχει η ολοκλήρωση της Ένωσης ε, δεν πρόκειται να προοδεύσουμε. Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης, ακούσαμε ότι μειώνεται πολύ η εμπιστοσύνη και όσον αφορά τις χώρες που ε, δεν ανήκουν στο ευρώ, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία, θα πρέπει να εξετάσουμε σε τι βαθμό μπορούμε να καλέσουμε τις χώρες αυτές να λογοδοτήσουμε. Ε, μια χώρα όπως ε, η, η Ουγγαρία έχει επιφυλάξει ως προς το ευρώ. Βλέπουμε άλλες χώρες όμως που έχουν προσχωρήσει στο ευρώ και που δεν ε, τηρούν τους κανόνες. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ευρωζώνη και δεν βλέπουμε διέξοδο. Επίσης, η προσφυγική κρίση έχει δείξει ότι υπάρχουν προκλήσεις στις οποίες δεν μπορούμε να δώσουμε γρήγορη και αποτελεσματική απάντηση. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω και τις προτάσεις μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται κάποιες ιστορίες επιτυχίας. Χρειάζεται από κοινού να βρούμε ε, σωστές ε, πρακτικές λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα απλώς να σας ζητήσω να ε, τηρείτε τα τέσσερα λεπτά. Η Πάρβαρα Σπινέλη από την Ιταλική ε, Βουλή. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κυρία Σπινέλη. Κύριε Πρόεδρε, να ε, καλωσορίσω τον κύριο Μόντι και τον κύριο Βιτορίνο και να τους ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις τους. Θα ήθελα να πω ότι ο όρος ε, πολυκρίση δεν με ε, πείθει. Πρόκειται για έναν όρο ο οποίος απλώς ε, ωρεοποιεί λίγο την πραγματικότητα. Εγώ θα τολμούσα να μιλήσω για μια αποτυχία. πρέπει να βγούμε από αυτή την αποτυχία, αλλά δεν πάβει να είναι αποτυχία. Ο κίνδυνος που διαβλέπω είναι να απαντήσουμε σε μια ευρύτατη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών, ε, προτείνοντας συνεχώς ε, τις ίδιες πολιτικές στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ο Βόλκαν Μούχα αποτελεί ε, η στιγμή της Μαρίας Αντουανέτας. Δηλαδή, υπάρχει μια στεναρή αντίδρυση απόρριψης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί στείνουμε να απαντούμε πάντα με τις ίδιες λύσεις. Η υπενθύμηση της υπόθεσης της Συμφωνίας ΣΥΤΑ μου φαίνεται εμβληματικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα ε, σημαίνουσα, διότι είναι αλήθεια ότι αφαιρώντας αρμεδιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά τις αφαιρούμε και την ομιμοποίηση. Αυτό το οποίο υποπτεύομαι είναι ότι αφαιρεώθηκαν αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπήρχε ήδη κρίση νομιμοποίησης. Δηλαδή, αυτή η μεικτή συμφωνία Εθνικών Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλεται σε μια κρίση νομιμοποίησης η οποία προϋπήρχε. Και θα συνοψίσω ε, με δύο λόγια μόνο αυτά, για αυτά τα οποία θεωρώ προτεραιότητα για να μπορέσει η, να υπάρξει αυτή η αξιοπρεπής Ευρώπη στην οποία αναφέρθηκε ο καθηγητής Μόντι, το πρώτο στοιχείο, η πρώτη προτεραιότητα είναι η δημοκρατικοποίηση και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη με ε, ισχυρά μέτρα δημοκρατικοποίησης, παραδείγματος χάρη με τους ίδιους πόρους. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, την έκθεση είναι θεμελιώδης οι πόροι για τις νέες λειτουργίες μας, ε, τα νέα καθήκοντά μας, αλλά κατά την άποψή μου θα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να υπενθυμίσουμε και την πτυχή της διαφάνειας ε, στη διαχείριση των ίδιων πόρων. Ε, πιστεύω μεταξύ άλλων ότι τα δημοψηφίσματα δεν είναι απαρατήτως μορφή μομφής και αν ζούμε συνεχώς με το φόβο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν θα κάνουμε αυτή τη δημοκρατικοποίηση. Κατά την άποψή μου, οι οικονομικές ε, ε κρίσεις θα οδηγήσουν και σε κοινωνικές συνέπειες, αλλά θα υπάρχουν και ε, πάρα πολύ σημαντικές ε, παράμετροι της κρίσης στα κοινωνικά ζητήματα. Τέταρτο σημείο, οι μεταρρυθμίσεις και η κοινωνική πτυχή. Αυτό σχετίζεται και σε αυτό που έλεγα για τη ΣΥΤΑ. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση έχει μια τάση να αφαιρεί πολλές εξουσίες, αρμοδιότητες και αποφάσεις από τους εθνικούς νομοθέτες. Αυτή είναι η άποψη που έχουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω είναι κάτι για τη συνθήκη. για τα σχέδια ή να συνεχίσουμε με αυτή τη συνθήκη ή να έχουμε μια νέα συνθήκη. Κατ' ουσίαν θα ήθελα να πω ότι μια συνθήκη που φιλοδοξεί ε, να είναι συνταγματική δεν είναι φτιαγμένη για να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, και ταχύτητα ε, κάποια πολιτική. Ο στόχος ενός συντάγματος δεν θα έπρεπε να είναι αυτός το Σύνταγμα υποδεικνύει προς να οργανώσουμε τη μορφή του κράτους, τις ισορροπίε μεταξύ των εξουσιών, τι υπηρεσίε μεταξύ εξουσιών και ο εξουσιών στο άλλο φάσμα και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και άμεση δημοκρατία, γιατί ε, την έχουν ανάγκη οι πολίτες την αμεσοδημοκρατία. Ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για τη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να αποπειραθούμε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, δεν έχω δυνατότητα να σα διακόπτω και δεν θα το ήθελα κιόλα. Γι' αυτό θα ήθελα να σα ζητήσω να τηρείτε τα αυτά τα 4 λεπτά χρόνου αγόρευση. Κύριο Κάσου. Λυπάμαι που ο κύριος Φερχόφστατ δεν είναι εδώ, γιατί πράγματι θα ήθελα να συζητήσω τις προτάσεις που, μαζί του τις προτάσεις που υποβάλλει. Εγώ έχω επισκεφθεί την Πρατισλάβα πολλές φορές τους τελευταίους μήνες. Και ήμουν από αυτούς που ζητούσα ε, στην ε, προκλητική εκστρατεία του Ηνωμένου Βασίλειου το Ηνωμένο Βασίλειο να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα που έχει οδηγήσει στην έλλειψη εμπιστοσύνη είναι το γεγονό ότι οι δημοκρατικέ διαδικασίε στην Ευρώπη δεν λειτουργήσαν. Ε, αυτός ήταν ο σεισμός. Έχουμε μία κατάσταση όπου η Ευρώπη κινείται προς όλο και μεγαλύτερη αστάθεια. Αυτό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ γεννήθηκα 10 Μαΐου του 40 και έζησα κάποια από αυτά τα, τα γεγονότα. Λοιπόν, τη δεκαετία του 50 και του 60 ε, μέχρι το 75 ε, υπήρχε η αίσθηση ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ε, σταθερότητα. Εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησα τη θητεία μου το 1984. Και διαπίστωσα όμω ότι τώρα πια, τότε πια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούσε πλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργούσε αστάθεια. Και βρισκόμαστε πλέον ενώπιον μια κρίση. η οποία έχει εξαπλωθεί παντού, θα τη δούμε και στην Ιταλία, έχει φτάσει στη Γαλλία, ε, στη Γερμανία, μέρος της κρίσης είναι και το προσφυγικό πρόβλημα. Επομένως, τι προσπαθώ να πω. Η ουσιαστική ερώτηση που αφορά τη δημοκρατία είναι πώς μπορούμε δημοκρατικά να συμφωνούμε και να επιλέγουμε στις κάλπες. Εγώ δεν συμφωνώ με εκείνους που θεωρούν δειλία ή έναν τρόπο να ξεφύγει κανεί από τι ευθύνε του στο δημοψήφισμα. Αντιθέτω, είναι ένα, θα, μια θαραλέα πράξη. Γιατί δίνει με τη δυνατότητα στου πολίτε να εκφραστούν και να καταγγείλουν πράγματα, όπω για παράδειγμα την ανεργία ή την αυξανόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα η οποία πλήττει τους πολίτες. Ε, και για να έρθω στο ζήτημα του Brexit. Κλείνοντας. Η διαδικασία του Brexit προχωράει. Δεν πρόκειται να συμβεί κανένα αρμαγεδόν. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκαν τα ε, αριθμητικά στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία του ε, Ηνωμένου Βασιλείου και διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί η αγοραστική ε, εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη του καταναλωτή μάλλον, οι, εξα... εξαγωγέ, οι επενδύσει. Έχουμε μεγάλε εταιρείε όπω η Google ή η Jaguar οι οποίε δημιουργούν θέσει εργασία. Ακόμα και η, και η Τράπεζα τη Βρετανία πηγαίνει καλύτερα. Χαίρομαι λοιπόν που καταφέραμε να φύγουμε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία απέτυχε να εκπληρώσει τις προσδοκίες που δημιούργησε και η οποία προσπαθεί να έρθει, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο αντιδημοκρατική, η οποία δεν εκπλήρωσε αυτό που το 1975, που ψηφίσαμε να ανταχθούμε, μας υποσχέθηκε. Γιατί το μόνο που μας, μας παρέμεινε αν παραμέναμε θα ήταν όλο και περισσότερες κρίσεις. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μαλότρα, από την Βουλή των Κοινοτήτων επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση τη σημερινή, μιας και είμαι μέλος της νέας ειδική Επιτροπής της Βουλής των Κοινοτήτων για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ενημερώσω επίσης ότι είμαι μέλος ε, ε, των εργατικών και έως πρόσφατα συμμετείχα και στην Επιτροπή για τα Οικονομικά. Ο Βίλιαμ, κύριος και εγώ μπορεί να διαφωνούμε. Εγώ υποστήριζα την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι επειδή πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέλεια. Αντιλαμβανόμαστε, αντιλαμβάνομαι ότι όταν υπάρχει ένας πολύπλοκος πολιτικός οργανισμός, αυτός θα χρειάζεται συνεχώς να εξελίσσεται, αλλά ζητούσαν την παραμονή μας και ε, ε, ε, υποστήριζαν την παραμονή μας επειδή πιστεύω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ωφεληθεί τα μάλα και επίσης επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει την ειρήνη στον, στην, στην Ευρώπη πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τέτοια πρωτοβουλία στον κόσμο, στην ιστορία. Τα ζητήματα αυτά δεν αναδείχθηκαν όπως έπρεπε στην εκστρατεία πριν το δημοψήφισμα. Και αυτό φάνηκε από το γεγονό ότι οι πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου είπαν ότι πριν το δημοψήφισμα δεν είχαν τι απαιτούμενε πληροφορίε, δεν γνώριζαν τι έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευημερία του και στην διασφάλιση τη ειρήνη. Είναι εύκολο να ζητάει από, από κάποιον να ψηφίσει να αποχωρήσει από έναν οργανισμό τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι έχει δημιουργήσει όλα του τα προβλήματα στη ζωή που αντιμετωπίζει αυτός ο πολίτης στη ζωή του ή επίσης ότι ευθύνεται αυτός ο οργανισμός για όλα τα προβλήματα που η χώρα θα έπρεπε να είχε λύσει. Επομένως οι συζητήσεις όπως αυτή που κάνουμε σήμερα θα συνεχιστούν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφορών εξουσιών και αρμοδιοτήτων και τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και για εμάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συζήτηση θα συνεχίσει γιατί θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάποια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ προσωπικά και πολλοί συνάδελφοι επιθυμούμε μια θετική ε, σχέση. Δεν πρόκειται να φύγουμε από την Ευρώπη. Είναι ε, ο φυσικός μας σύνοχος, σύμμαχος οι ευρωπαϊκές ε, χώρες. Επομένως η σχέση μας μαζί τους θα πρέπει να συνεχίσει να είναι θετική τα θέματα αυτά φυσικά τα συζητώ με τους πολίτες ε, στη χώρα μου, εκείνους που, που εκπροσωπώ και φυσικά οι Βρετανοί πολίτες ε, ανησυχούν. Δεν ισχύει μόνο αυτό που ε, ακούστηκε από τον συνάδελφο, δηλαδή το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία τα οικονομικά πηγαίνουν καλύτερα, υπήρχαν και αρνητικοί δείκτες. Όλο και περισσότερο νέοι άνθρωποι λένε ότι φοβούνται την ανεργία και ότι δεν βρίσκουν τις δουλειές που έβρισκαν στο παρελθόν όλη η συζήτηση που είχαμε το πρωί σε σχέση με τις εξεταστικές επιτροπές και την, τη συζήτηση που έχουμε τώρα μου δείχνει ότι πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο πώς θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε όλοι μαζί ως έθνος και πώς θα συνεργαζόμαστε. Ε, και θεωρώ ότι ένας από τους ρόλους που θα πρέπει να παίξει η Ειδική Επιτροπή για τον Brexit ε, να εξετάσει τα, τους κινδύνους που τίθενται και τις ευκαιρίες που ανοίγονται, αλλά ε, επίσης να ελέγξει την κυβέρνησή μας, τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί, αλλά επίσης να σκεφτούμε ποιες μεταβατικές ρυθμίσεις θα χρειαστούν, οι οποίες σίγουρα θα είναι περίπλοκες αλλά θα είναι αναγκαίες. Κλείνοντας, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις ότι η συζήτηση συνεχίζεται και είναι περίπλοκη. Για παράδειγμα, μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούμε απέναντι στην ελευθερία μετακίνησης προσώπων μετά το Brexit, εάν θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και τύπου έλεγχοι. Και πιστεύω, κλείνοντας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει ενωμένη να προχωράει προς το στο κοινό της μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται αλλαγή των συνθήκων. Ο κύριος Κάζ αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία δεν ε, αναφέρεται μόνο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών, αλλά επίση και στην εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων από τη μια και των κρατών μελών από την άλλη. Δεν πιστεύω ότι η ορθή απάντηση είναι η όλο και περισσότερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων. Με ανησυχεί το γεγονό ότι διαπιστώνω όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν άλλον τρόπο λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πώς να λειτουργεί. Εγώ πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να το αφήσουμε να επιλέξει μόνος του, μόνο του πώς θα λειτουργεί. Οι διερμηνεία ζητούν να κλείσει το μικρόφωνο της Πρόεδρος γιατί υπήρχε θόρυβος. Ε, η σταθερότητα των ε, δημοσίων οικονομικών έχει πολύ μεγάλη σημασία Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η ενιαία αγορά ε, σκοντάφτει και σε διάφορα εσωτερικά εμπόδια. Ένα τρίτο θέμα εξίσου σημαντικό είναι η διαφάνεια. Και η έκθεση γίγκα για το θέμα αυτό θα πρέπει να, για το θέμα της διαφάνειας πρέπει να τη λάβουμε πολύ σημαντικά. Σοβαρά. Υπόψη μας. Έρχομαι τώρα στο θέμα των συνθήκων. Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη διαδικασία, η διαδικασία της επικύρωσης μιας διεθνούς συνθήκης σε οποιαδήποτε χώρα. Πάντα χρειάζεται ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της χώρας, πάντα χρειάζεται σε κάποιες χώρες δημοψήφισμα, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση σε μια ιστορική στιγμή. Και πρέπει όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε τις πολύπλευρες κρίσεις που έχουν πλήξει τις χώρες μας. Συμφωνώ ε, σχεδόν σε όλα με αυτά που είπε ο κύριος Μόντι. κυρίως ότι θα πρέπει ουσιαστικά να ασχοληθούμε με το ζήτημα το πολιτικό και το πολιτισμικό. Είναι σημαντικό για εμάς που είμαστε από τα ιδρυτικά κρατημέλη, αλλά είναι σημαντικό και για όλα τα άλλα κρατημέλη. Ποιος είναι ο ρόλος των ε, κοινοβουλίων στην ε, επίλυση αυτών των προβλημάτων. Είναι ουσιαστικότατος. μιας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις οι οποίες προέρχονται και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι κοινοί μας στόχοι, ποια είναι οι κοινέ επιδιώξεις που μας κάνουν να συνεχίσουμε να, συνεχίζουμε να επιθυμούμε να είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε και ο κύριος Μπρόκ στο προσεχές ε, δημοψήφισμα στην Ιταλία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την κυβερνησιμότητα της Ιταλίας που τίθεται στους Ιταλούς πολίτες. δεν πρόκειται ε, συνεχίζει να υφίσταται τη διάκριση μεταξύ της ε, ε, άμεσης έκφρασης της άποψης των πολιτών και της διακυβέρνησης. Και κλείνοντας, για το ζήτημα της επικύρωσης της ΣΥΤΑ και μας, μας απασχόλησε το θέμα του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων σε μεικτές συμφωνίες όπως αυτή όπου υπάρχουν συντρέχουσες αρμοδιότητες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών. Εδώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν και εκείνα λόγο και να συμμετέχουν στη διαδικασία επικύρωσης. Πρόκειται για διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Είναι ε, ε, απολύτως απαραίτητο τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν να, να τους επιτρέπεται να συμμετέχουν. Γιατί ορισμένες φορές μπορεί να βρισκόμαστε στην πλειοψηφία, να συμφωνούμε με την άποψη της πλειοψηφίας, όμως σε άλλες περιπτώσεις θα βρισκόμαστε με την πλευρά της μειοψηφίας και αυτά πρέπει να γίνεται σεβαστό. Όσον αφορά τα δημοψηφίσματα, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλέ φορέ για να αποσταλεί ένα μήνυμα διαμαρτυρία από του πολίτε απέναντι στο κατεστημένο που θεωρούν ότι δεν του εκφράζει πια. Το άρθρο 138 του Ιταλικού Συντάγματος προβλέπει ότι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία δύο τρίτων για μια συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα ε, διεξάγεται δημοψήφισμα. Και αυτό συμβαίνει ε, τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να είσαστε πιο σύντομοι. Ο κύριο Αντρώνη Ασούπαλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, ποιοι θα σας αναδημορφώσουν, η Ευρώπη ή τα κράτη-μέλη. Σε ποιον ανήκει το εγχείρημά σας. Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα. Σήμερα όμως δεν νομίζω ότι βρήκαμε απάντηση σε αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναστούμε την απάντηση. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση που παρουσίασε ο αγαπητός μου φίλος Έλμαρ και ε, η αξιολογή συνάδελφός του. Η έκθεση αυτή οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση σε Ευρώπη πολλών ε, ταχυτήτων, ε, πιο πιθανό όμω να μην οδηγεί καθόλου στην Ευρώπη. Ε, μερικοί θα έλεγαν ότι τα μέτρα που προτείνονται δεν αποτελούν μέσο για την θεσμική βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για τη διάλυσή της. Η συγκέντρωση εξουσιών, το να εγκαταλείψουμε την ομοφωνία είναι αρκετά προκλητικές προτάσεις οι οποίες ε, ήδη ε, έχουν ε, φανεί καταστροφικές. Ας θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν. Μέσως πριν το δημοψήφισμα, οι ηγέτες ήθελαν εμβάθυνση της Αμυντικής Ένωσης και αναθεώρηση του εκλογικού νόμου και είδαμε την αντίδραση του κοινού. Μπορεί να είναι ρητορικό το ερώτημα, μπορεί όμως και κάποιος να έχει κάποια απάντηση. Γιατί ε, δίδονται τέτοιες φυγοκεντρικές προτάσεις από πλευράς των Βρυξελών. Ε, τέτοιες κινήσεις αυτή τη στιγμή θα οδηγήσουν μόνο σε ανεπιθύμητες ε, συνέπειες. Το να δώσουμε περισσότερες εξουσίες ε, στο κεντρικό επίπεδο, ε, να μην θίξουμε όμως ε, τις συνθήκες, δεν είναι κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση. Δεν νομίζω θα πρέπει να φοβηθούμε τα πιθανά σενάρια για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητήσουμε ανοιχτά τα υπέρ και τα κατά. Πολλοί αντικειμενικοί παράγοντες δείχνουν ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να γίνει περισσότερο ακουστή η φωνή τους. Επίσης, ε, το κράτος έθνος είναι ο εγγυητής της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, ε, ο μόνος τρόπος να λύσουμε αυτό το θεσμικό πατ είναι ε, να έχουμε πάντα ομοφωνία, να μην έχουμε ψηφοφορίες με ειδική πλειοψηφία. Ε, στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε το τέλειο σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο να πετυχεί κανεί την ομοφωνία, αλλά αυτή είναι η δουλειά μα ως πολιτική. Η ειδική πλειοψηφία οδηγεί σε περισσότερες διαμάχες και ε, έχει ε, μέσα τις, τις διαμάχες και τις αντιθέσεις. Φοβάμαι ότι αν ε, ακολουθήσουμε την ε, ίδια παλαιά οδό θα οδηγηθούμε σε περισσότερες εξόδους. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Τριανταφύλου, παρακαλώ, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Η κορύφωση της ε, προσφυγικής κρίσης με τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μια σειρά αλλεπάλληλων κρίσεων, δοκίμασαν και δοκιμάζουν ως σήμερα την εντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέτοιμη, αμήχανη και αναποτελεσματικής ως προς τη διαχείρισή τους. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί μια σειρά από χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, να μπαίνουν στο άρμα της χρεομηχανής και το χρέος να γίνεται εργαλείο χειραγώγηση των λαών που παρακολουθεί την ανεργία να καλπάζει, τη λιτότητα να απλώνεται, τη διαφάνεια να αναζητείται, που παρακολουθεί βασικέ τις επιλογές και θεσμίσει όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να μην λειτουργεί ενισχυτικά στην παραγωγή, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περαιτέρω ελλημάτων, που παρακολουθεί τη σταδιακή αποδόμησή της. Είναι ώρα για μια εκ νέου διαμόρφωση της συλλογική μας συνείδησης και αποτελεί αναγκαιότητα και πρόκληση συνάμα η αναβάπτιση των ευρωπαϊκών ιδεών, της ελευθερίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ισοπολιτείας, των ανθρωπίνων, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τη κοινωνική συνοχή του σεβασμού της διαφορετικότητα. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη σχέση συλλογικού ατομικού, τέτοια που θα αποκαθιστά τη σημασία του συλλογικού στα μάτια του κόσμου, των λαών. Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα έχουν ως στόχο την εμβάθυνση τη δημοκρατία, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου, τη δίκαιη ανάπτυξη με οικολογικό πρόσημο. Θα έχουν ως στόχο την ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας, την αποφυγή της μετατροπής της Ευρώπης σε Ευρώπη φρούριο, σε Ένωση φρούριο, που θα επιλύουν την προσφυγική κρίση όχι μόνο με όρους αλληλεγγύης και φιλοξενίας, αλλά με ουσιαστικές πρωτοβουλίες για ειρηνική επίλυση των διαφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, της Συρίας, με καταδίκη των πολεμικών των τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και με καταδίκη της εξαγωγής δημοκρατίας στην οποία πήραν και παίρνουν μέρος πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και βέβαια, με λύση του Κυπριακού. Σήμερα υπάρχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεχόμαστε όλες οι υπόλοιπες χώρες την εισβολή και κατοχή. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να πούμε συγκεκριμένε προτάσει. Για παράδειγμα, οι προτάσει που διατυπώνονται στη διακήρυξη των Αθηνών. Μια πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με στόχο την προώθηση του διαλόγου για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για τη λήψη γενναιότερων αποφάσεων στο πλαίσιο τη Ένωση, τέτοιε αποφάσει που έχουν ανάγκη όλοι οι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του στο ευρωπαϊκό όραμα. Ενδεικτικά αναφέρω στον οικονομικό τομέα διπλασιασμό της χρηματοδοτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προώθηση επενδυτικών σχεδίων σε κράτη-μέλη με υψηλή ανεργία και διασυνοριακά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, των πρακτικών φορολογικού και κοινωνικού ντάπινγκ. Για το μεταναστευτικό, υιοθέτηση μιας συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα περιλαμβάνει ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με τη μετεγκατάσταση. Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης και των δυνατοτήτων κινητικότητας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράνομης μετανάστευσης. Ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και με τις αφρικανικές χώρες. Τέλος, δύο σημεία. Υπάρχει αδύρυτη ανάγκη επαναπροσδιορισμού και επανανοηματοδότησης τη έννοια της λογοδοσία η νομιμοποίηση των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου είναι υπαρκτή, αλλά όχι παντοτινή. Και οι λαοί δεν είναι άβουλο σώμα που περιμένουν από τις ειδήσει να μάθουν τις θεσμίσεις. Τις βιώνουν. Και ένα τελευταίο για το δημοψήφισμα. Η κάθε χώρα έχει τη δική της εμπειρία. Μπορεί ωστόσο ένα δημοψήφισμα να μεταμορφώσει τον κόσμο σε λαό. Τότε ενδυναμώνει μια συλλογικότητα, μια πολιτική εξουσία, μια κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Mm, σας ευχαριστώ πολύ. Από την Πολωνία. Ο κύριος Βιασόσκη. Słuchałem głosu sprawozdawców, e, żeby dokładnie wych... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Διάβασα με προσοχή την ε, πρόταση του ε, εισηγητή και τους συναδέλφους. Πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσουμε στο εξής ότι δεν αρκεί να ακούμε ο ένας τις απόψεις του άλλου εδώ στην αίθουσα μεταξύ μελών κοινοβουλίων. Πρέπει να βγούμε προς τα έξω στους πολίτες να ακούσουμε τη δικιά τους άποψη. Γιατί βεβαίως ίσως κάποιοι συνάδελφοι να με πείσουν σήμερα εδώ. Αλλά πώς θα γυρίσω εγώ στην Πολωνία και θα πείσω τους πολίτες μου ότι ε, λάθος κάνουν, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Όταν γνωρίζω ότι οι πολίτες στην Πολωνία, η πλειοψηφία τους δεν επιθυμεί μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Αυτό που θα ήθελαν η, πλειονότητα των Ευρωπαϊκών πολιτών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ισχυρή, να εγγυάται την ασφάλειά τους, να είναι ορθολογική και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τις ίδιες παλιές απαντήσεις στα νέα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι γνωστό ότι αμφιβολίες και ανησυχίες για τον, την πορεία που έχει αρχίσει να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν εκφραστεί ήδη από τις ψηφοφορίες που γίνανε για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Και τότε οι ελίτ δεν άκουσαν τους πολίτες. Δεν βρήκαν μια σωστή ε, απάντηση να δώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν περαιτέρω ολοκλήρωση. Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνταγή. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε, να νομίζουμε όταν οι πολίτες μας το λένε με τόσους διαφορετικούς τρόπους ότι η λύση είναι η περισσότερη ολοκλήρωση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια, μια κοινή, Ευρώπη. Όχι, εμεί θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να σέβεται και να βασίζεται πάνω στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών τη. Συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ. Θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ε, διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύγχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επιδείξει τη διαφάνεια που θα έπρεπε. και εμείς που βρισκόμαστε στα εθνικά κοινοβούλια το έχουμε διαπιστώσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κίτρινη κάρτα που έβγαλαν 11 εθνικά κοινοβούλια για την ε, ε, οδηγία για το κοινωνικό ντάμπινγκ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε ανακοινώσεις, τις δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της και μετά απλώ ζητάει από τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται καν από τη συνθήκη να μας φέρνει πρωτετελεσμένων γεγονότων η Επιτροπή. Επομένως, στο ερώτημα του κυρίου Μπροκ, μήπως θα έπρεπε α, η εφαρμογή των συνθήκων να διευρυνθεί. Να σας υπενθυμίσω κύριε Μπρόκο ότι ήταν το γερμανικό συνταγματικό δικαστηρίο το οποίο ε, είπε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να κυκλώνουν συνθήκες και το είχε ε, διευκρινίσει αυτό με την ευκαιρία της συνθήκης του Μάστριχτ. Όπως συμβαίνει όταν κανείς προσπαθεί να ακολουθήσει συνταγή, έχει σημασία η λεπτομέρεια. Έχουν σημασία όλα τα μπαχαρικά. Δεν αρκεί να φτιάξουμε κάτι στο περίπου. Αυτό δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νόρτβις, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ποια είναι η νομιμοποίηση αυτού του καταπληκτικού εγχειρήματος της Ευρώπη Και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε πώς μπορούμε να ενεργήσουμε βραχυπρόθεσμα και πώς μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε στα σοβαρά την δημοκρατία και τη διαφάνεια. Διότι όταν βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες με την Ευρώπη, πολύ συχνά οφείλονται στην έλλειψη διαφάνειας. Είναι αποφασιστικής σημασίας να έχουμε διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα. Με εξέπληξε που άκουσα τον κύριο Μόντι να μιλάει για την επικύρωση ε, διαφόρων συμφωνιών. Εάν δηλαδή ε, κάποιος ε, δεν μπορεί να... Αν υπάρχει μια πρόταση που θα πρέπει να πει ναι ή όχι σε όλη την πρόταση. Αλλά έτσι δημιουργούμε συγκρούσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την μη επικύρωση από κάποια κοινοβούλια. Θα πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον. Πριν λίγες εβδομάδες είδαμε το τι έγινε ε, όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας ΣΥΤΑ που ακούσαμε ε, διάφορες προειδοποιήσεις από διάφορα κρατημέλη και τελικά είδαμε ε, την Βαλονία μόνο να να ε, εμφανίζεται αντίθετη σε τόσους ε, ισχυρού. Θα πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Oh, uh, Ήσασταν σύντομο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ο μιλητής, ο κύριο Γιώνα Γκούναρσον. Σα ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα συμφωνήσω με τον Έλμπαρ Μπροκ που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει αυτά που έχουμε συμφωνήσει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, κάνουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς βλέπουμε να μην λειτουργεί το σύστημα αυτό. Και εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Η έλλειψη αλληλεγγύης που βλέπουμε ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποτελεί το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί την αντίθεση και όχι το αν λειτουργούν τα θεσμικά όργανα με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Σίγουρα είναι και αυτό σημαντικό. Είναι σημαντικό να λειτουργεί σωστά το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτά που συμφωνούμε δεν εφαρμόζονται. Έχουμε σαφή παραδείγματα, όπως για παράδειγμα κατά την μεταναστευτική κρίση. Αυτό είναι κάτι που διακυβεύει την ε, εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη ευθύνη, έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς, ε, τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις στις πρωτεύουσε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά το σύστημα εάν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά. Εάν δεν υπάρχει αλληλεγγύη, το σύστημα θα καταρρεύσει. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί με τροποποίηση της ε, συνθήκης. Αυτό έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Εμάς ε, που καθόμαστε εδώ στο τραπέζι των συζητήσεων. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, το σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, πριν από έξι χρόνια αποκτήσαμε ένα μέσω ε, ε, στα κοινοβούλια να εξετάζουμε κατά πόσο οι προτάσεις ε, συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. Δυστυχώς τα, ευρωπαϊκό, τα, τα εθνικά κοινοβούλια ελάχιστα έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο ελάχιστα κοινοβούλια εξετάζουν ε, το κατά πόσο συνάδουν οι προτάσεις ε, με την αρχή της επικουρικότητας. Ε, εάν λοιπόν δεν πάρουμε στα σοβαρά τα δικά μας καθήκοντα, τις δικές μας αρμοδιότητες, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει κανείς άλλος. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στους συναδέρφους στα Εθνικά Κοινοβούλια. Πάρτε στα σοβαρά το ρόλο σας, επιστρέψτε στο κοινοβούλιο σας, ε, απαιτήστε ε, την ε, λογοδοσία από τις κυβερνήσεις σας, διότι αυτές εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να περάσω στα μέλη του πάνελ και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μόντι κάποιες πρώτες αντιδράσεις και μετά οι Μερτσέτες και μετά ο Έλμαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία παρατήρηση θα κάνω μόνο που είναι η βασική μου αντίδραση σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σαφές, γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται σε ε, μια βαθιά κρίσιμη κατάσταση είναι ενδιαφέρον πως ε, πολλοί τείνουν ε, να αποδίδουν την μεγάλη δυσλειτουργικότητα της Ευρώπης ε, πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως επισημαίνουμε τη σημασία της δημοκρατίας και στο να εισακούγεται η φωνή των πολιτών και αν δεν έδωσα την εντύπωση ότι με ενδιαφέρει να διορθώσω αλλά είναι σαν να ρίχνουμε το φταίξιμο για όλα όσα δεν λειτουργούν στην Ευρώπη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ την χάνει να πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι τα εθνικά πολιτικά συστήματά μας τα οποία είναι όλο ένα και πιο δυσλειτουργικά και αντιμετωπίζουν κρίση και έχουν κρίση νομιμοποίησης. Είμαι όπως πολλοί από εσά εδώ μέλος ενός Εθνικού Κοινοβουλίου. Είμαι μέλος της Ιταλικής Γερουσίας. Και σε όλους αρέσουν οι δημοκρατία μας και όλοι ελπίζουμε να παραμείνουμε δημοκρατικοί. Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η λειτουργία των εθνικών πολιτικών μας συστημάτων είναι κατά βάση ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε τέτοια κατάσταση. Με δύο λόγια. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε εθνικά πολιτικά συστήματα στα οποία υπήρχε ηγεσία. Αυτό αυτή τη στιγμή με τα εθνικά πολιτικά συστήματα τα οποία ολοένα και περισσότερο ε, καταλαμβάνονται από βραχυπρόθεσμα πράγματα. Ε, απλώς εξετάζουν ε, ε πώς να εκλεγεί κάποιος ε, και μόλις συσταθεί η κυβέρνηση πώς να επανεκλεγούν. Επομένως, πολύ βραχυπρόθεσμος ορίζοντας η έλλειψη οποιασδήποτε προσοχής στο μακροπρόθεσμο. Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Κίνας στην πραγματικότητα, κάτι το οποίο δεν είναι καλό για την Ευρώπη. Αλλά αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή ισχύει και σε μεγάλο βαθμό για την περίπτωση των ΗΠΑ. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η εξέλιξη της πολιτικής διαδικασίας σε κάθε μία από τις χώρες μας είναι αυτή η οποία είναι όλο ένα και πιο ασύμβατη με την ε, ολοκλήρωση. Μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εκτός και αν δώσουμε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Και φυσικά ε, θα πρέπει να δούμε και τα διδάγματα της ιστορίας για άλλη μια φορά. Χωρίς ολοκλήρωση, χωρίς κάποιες μορφές ολοκλήρωση, όχι αιμονική ολοκλήρωση, αλλά χωρίς ολοκλήρωση στην Ευρώπη έχουμε πόλεμο. Τελεία και παύλα. Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και από τους ηγέτες τους να δημιουργήσουν ε, ένα κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι και προς τα εθνικό συμφέρον. Τώρα γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Το Brexit και αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργό Κάμερον, είναι στον υπερθετικό βαθμό, είναι αυτό το οποίο κάνουν οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Δρούν απλώς και μόνο για το δικό τους πολιτικό κόμμα και τα προσωπικά τους συμφέροντα, ούτε καν για την χώρα τους. Εγώ είχα την τιμή να είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακόμα και η φύση ε, με, τον οποίο, ε, με την οποία ε, δεχόμαστε τις δημοκρατίες μας, όχι με αυτή την αιμονή, όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές, γιατί οι επόμενες εκλογές είναι, δεν, δεν είναι σε ορίζοντα ενός-δύο ετών, υπάρχει η επόμενη σπιχομομέτρηση που λαμβάνουν υπόψη τους οι πολιτικοί. Και έχουμε 28 άνδρες και γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που παριστάνουν ότι αποφασίζουν για την Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας από αυτούς προσπαθεί να προωθήσει τις δικές του τις θέσεις. Και το γεγονός ότι το Brexit μας προέκυψε και ο κύριος Κάμερον και λυπάμαι πολύ διότι είχα εξαιρετικές σχέσεις μαζί του ε, πλήρωσε ένα τόσο με βαρύ πολιτικό τίμημα κρούει λίγο τον κόδωνα του κινδύνου για τους άλλους πολιτικούς ηγέτες για να μην είναι τόσο κοινικοί πιστεύω ότι εάν δεν αλλάξουμε εμεί ως πολίτες, δεν επιδείξουμε πιο υπεύθυνη συμπεριφορά ε, για τα δικά μας εθνικά πολιτικά συστήματα και τους δικούς μας εθνικούς ηγέτες στην εθνική, η διεθνή ολοκλήρωση, θα είναι όλο ένα και πιο απροσπέλαστη. Και θα δούμε ότι αυτό θα είναι εις βάρος της Ευρώπης και στη συνέχεια αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσείς, ε, δηλαδή ναι με να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη αλλά χωρίς ολοκλήρωση, δυστυχώς, είναι οξύμορο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη μετά από 10 χρόνια ε, θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρία σε ένα κράτος μέλος. Μην πιστέψουμε ότι αν κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχη ε, με το εξαιρετικό παιχνίδι της εθνικής μας δημοκρατίας θα λειτουργήσει. Γιατί η δυσλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι οι εθνικές μας δημοκρατίες δεν είναι πλέον αρκετά σοβαρές ώστε να υποστηρίξουν τη διαδικασία της ολοκλήρωσης που είναι η μόνη εναλλακτική λύση για τον πόλεμο. Συγγνώμη αν ήμουν λιγάκι όμως. Νομίζω ότι από καιρούς καιρών χρειαζόμαστε λίγο πιο ε, ε, γλώσσα. Μεσέντες, Έλμαρ, θέλετε να απαντήσετε. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος. Η Μερσέντεν μου είπε ότι πρέπει να αρχίσω εγώ, λέει ο κύριος Σπρόκ. Καταρχά η κρίση νομοποίησης τη δημοκρατία δεν είναι αποκλαστικά ευρωπαϊκή. Αυτό το βλέπουμε και στα κράτη-μέλη. Ε, μην ε, κατηγορείτε μόνο την Ευρώπη. Αυτό ε, είναι πολύ εύκολος τρόπος. Όταν ε, βλέπω την κατάσταση στα κράτη-μέλη, βλέπω ότι είναι η ίδια με την Ευρώπη. Ε, μην πέσετε θύματα του λαϊκισμού, δεν φταίει μόνο η Ευρώπη. Δεύτερον, ε, οι αρμοδιότητες ανοίγουν στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη εκχωρούν ε, τις αρμοδιότητες και μπορούν να τις ε, πάρουν πίσω. Δεν τις πήρε τις αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις έδωσαν τα κράτη-μέλη. Και στην έκθεση δεν ζητάμε νέες αρμοδιότητες. Επίσης, Θα παρακολούσα ε, τον Λούκα να μα αφήσει να κάνουμε εμεί τη δουλειά μα, όπω και εμεί σα αφήνουμε να ασχοληθείτε μόνοι σα με τον Brexit. Και ας πάρουμε παράδειγμα την Βρετανική κυβέρνηση. Πριν το Brexit ε, έγινε μία μελέτη σχετικά με το ποιες ε, αρμοδιότητες ε, θα πρέπει να ξαναπάρει πίσω το κράτος ε, και η απάντηση ήταν μηδέν, καμία. Άρα δεν είναι θέμα αρμοδιοτήτων, είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τις αρμοδιότητες. Και μπορεί πάντα να συζητάει κανείς εάν έγινε με σωστό τρόπο ή όχι. Άλλωστε δεν άκουσα ούτε εδώ καμία πρόταση για το ποιες αρμοδιότητες θα πρέπει να πάρουν πίσω τα κράτη-μέλη. Κανένας σήμερα δεν υπέβαλε τέτοια πρόταση. Μιλάμε δηλαδή για το πώς ε, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ε, τις αρμοδιότητες ε, που έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δίνετε αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώστε τις και εργαλεία για να τις ασκήσει. Ε, εδώ και πολύ καιρό τα, ε, προτάθηκε μια ευρωπαϊκή ε, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη αρνήθηκαν. Τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση, τα κράτη-μέλη απορρίπτουν. Τώρα έχουμε τη διαδικασία της Μπρατισλάβα με καλύτερες ε, δομές. 200 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουν τα κράτη-μέλη για την άμυνα τους ε, με ελάχιστο αποτέλεσμα. Ε, δίνουμε περισσότερα χρήματα στην άμυνα από ότι η Ρωσία. Έχουμε περισσότερους στρατιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με ελάχιστο αποτέλεσμα. Ε, και στη δική μου χώρα δεν είναι καλά τα πράγματα. 200 δισεκατομμύρια σπαταλάμε ε, λόγω έλλειψης ε, συνεννόησης. Και δεν μπορούμε καν να αγγιηθούμε την ασφάλεια της Πολωνίας. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλά τέτοια παραδείγματα. Ο Μαριομόντι το γνωρίζει καλύτερα από μένα διότι ήταν και επίτροπος, ε, ήταν και επικεφαλής της κυβέρνησής του. δεν ε, δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εργαλεία που χρειάζεται για να ε, κάνει τη δουλειά της. Δεν θέλουμε λοιπόν περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε καλύτερη Ευρώπη στο πλαίσιο των δεδομένων αρμοδιοτήτων. Ε, μην δίνετε αρμοδιότητες χωρίς να δώσετε τα εργαλεία για να λύσει τα προβλήματα. Ε, αυτό είναι θέμα απλής λογικής, διανοητικής καθαρότητας. Η Δανία είναι παράδειγμα. Τα... Η διαμαρτυρία της Βαλονίας ε, δεν είχε στραφεί κατά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κατά της πλειοψηφίας του Βελγίου και κατά των άλλων 27 κρατών μελών ήταν. Διότι τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια ήθελαν τη συμφωνία ΣΥΤΑ και νομίζω ότι τέτοια προβλήματα θα πρέπει να λύνουμε αν λέμε ότι οι ενέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διότι ε, κανένα κράτος μέλος ε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τότε θα πρέπει να δίνουμε τα απαραίτητα εργαλεία για στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπω θέλει το Λουξεμβούργο και η Μάλτα ε, να διαπραγματευτούν μόνοι του την επόμενη εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Το ίδιο ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θέλετε να διαπραγματευτείτε εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, σαν να είσαστε το 52ο ε, κράτος μέλος. νομίζετε ότι τα μεγέθη είναι τέτοια που θα σας δουν σαν ίσο εταίρο. Η επικουρικότητα είναι Επίσης, ε, σημαντικό να τηρείται, αποτελεί σημαντική υποχρέωση. Πρέπει όμως να υπάρχει και αλληλεγγύη και είναι πολύ δύσκολος ο ορισμός της αλληλεγγύης. Μεγάλες χώρες ε, έχουν άλλες προτεραιότητες από ότι οι μικρές. Ε, γενικά οι χώρες μεταξύ τους έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Ε, συμμετείχα τότε που δημιουργήσαμε την πορτοκαλί κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει επαρκής αριθμός εθνικών κοινοβουλίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να δώσουν τέλος στην νομοθετική διαδικασία χωρίς να εμπλακεί η Κομισιόν. για να λύσουμε το πρόβλημα της επικουρικότητας. Στην έκθεσή μας προτείνουμε οι προϋποθέσεις για τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια για τα εθνικά κοινοβούλια για να ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό να βελτιωθούν. Προσφέρουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βελτιωθούν ε, οι προϋποθέσεις και πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε και δεν ε, μιλάμε για περισσότερη ολοκλήρωση, μιλάμε για αποτελεσματική εφαρμογή και δημοκρατική νομιμοποίηση όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι εθνικές κυβερνήσεις να ξεφεύγουν από τις ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες τους. Το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάτι, όπως λέγεται συχνά, είναι λάθος. Ε, καμία νομοθεσία δεν ε, εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν λοιπόν οι εθνικές κυβερνήσεις κάνουν σαν να μην είχαν εμπλακεί καθόλου στην υπόθεση, αυτό είναι λάθος. Αυτό λοιπόν ε, είναι το θέμα κλειδί της διαφάνειας. όταν βλέπω τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν και από ποιον μπορούν ε, να λυθούν, καταλήγω πολύ σύντομα σε ένα συμπέρασμα. Λέμε ότι όλοι επικρίνουν την Ευρώπη. Ε, έτσι γίνεται αντιληπτή η Ευρώπη, αλλά χάρη και της σταθερότητας ε, στα κράτη ή μέλη να σκεφτόμαστε λύσεις όπως κάνουν και οι πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ η Mercedes. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν σας άκουγα σκεφτόμουν να αυτό που είπε πριν από λίγο καιρό ο γερμανός φιλόσοφος Άμπερμας, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη ή θα καταφέρει να παραμείνει ενωμένη ή θα βγει από τη μελλοντική ιστορία του κόσμου. Η εντύπωσή μου είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία έκανε ήδη την επιλογή της να αποχωρήσει από τη μελλοντική ιστορία του κόσμου. Βεβαίως εμείς μπορούμε όλοι μαζί να αναλάβουμε την ίδια ευθύνη. Να ε, βγούμε βαθμιδών με τη μία χώρα μετά την άλλη, η οποία θα κάνει την έξοδό τη ε, με τη σειρά τους ή θα την προτείνει. Ε, και έτσι θα προσπαθήσει να ε, διαλώσει, διαλύσει την νομιμοποίηση που δημιουργήσαμε μετά από περίπου 60 χρόνια πλέον. Ε, θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω, όπως υπενθύμησε και ο συνάδελφος Μπροκ, στην ιστορία κάθε δημοκρατίας Μόνο ένας είναι ο τρόπος για να εγγυηθούμε το σεβασμό της διάθεσης των πολιτών ε, ε, σε μια ένωση ε, Αυτό είμαστε. Αν διαβάσετε τις συνθήκες, αυτό είμαστε. Είμαστε σχεδόν ομοσπονδία. Και επομένως θα πρέπει να εγγυηθούμε μία μέθοδο λήψης αποφάσεων που θα σέβεται την πλειοψηφία των πολιτών αυτής της Ένωσης και την πλειοψηφία των κρατών. Και αυτό κατ' ουσίαν είναι η μέθοδος που προβλέπουν οι συνθήκες και τώρα. Η πλειοψηφία των πολιτών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με μία ε, μειούμενη αναλογικότητα μεν, αλλά εκπροσωπεί τους πολίτες και υπάρχει και εκπροσώπηση των πολιτών που είναι η ειδική πλειοψηφία. Χωρί αυτό, μία ένωση η οποία πρέπει να πάρει πάρα πολλέ αποφάσει, διότι αυτές οι αρμοδιότητες, όπως υπενθύμησε ο συνάδελφος Μπρόκ, υπάρχουν. Ε, δημιουργήθηκαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με κύρωση από τα κοινοβούλια αλλά και με δημοψηφίσματα όπου προβλέπονται. Αυτές οι αρμοδιότητες λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουν να ασκηθούν διότι το γεγονός ότι δεν ασκεί κάποιος τις αρμοδιότητές του εγκαίρως με την ταχύτητα και την απαιτούμενη ποιότητα ε, ε, που ε, σημαίνει ότι ε, χάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αδύνατη η αγαστή της λειτουργία. Ε, Δυστυχώ δεν είχαμε εδώ και τον συνάδελφο Φερχόφστατ για να μιλήσουμε για τα κενά του συστήματος και τις δυνατότητες να, να βελτιώσουμε και να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτά τα οποία κάναμε όμως όλοι μα και εγώ ξεκινώ από την προϋπόθεση ότι το κάθε ένα από τα κράτη σα και τα κοινοβούλια σα, εσεί ή οι συνάδελφοί σα όταν δεν ήσασταν εσεί, έχουν ήδη κυρώσει. Αυτή λοιπόν είναι μια εξουσία που διαθέτει ήδη η οι συναδελφοι σα οταν δεν ησασταν εσει εχουν ηδη κυρωσει αυτη λοιπον ειναι μια εξουσια που διαθετει ηδη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν την, αρκεί, ε, την ασκεί με σαφή, διαφανό, δημοκρατικό τρόπο. Η πλειοψηφία δεν είναι δημοκρατία. Η ομοφωνία, συγγνώμη, δεν είναι δημοκρατία. Η ομοφωνία είναι μπλοκάρισμα, δυναμία λειτουργία. Και η συνήθεια, ακόμα και όταν οι συνθήκε προβλέπουν ε, σταθμισμένη πλειοψηφία, η συνήθεια να ψηφίζουμε συνέχεια ομόφωνα οδηγεί σε μπλοκάρισμα και σε συνεχή έκρηξη των ε, εθνικών συμφερόντων ε, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Προσοχή! Τα εθνικά συμφέροντα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αν είναι να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε μαζί. Πολλό δε μάλλον και τα μικρότερα κράτη-μέλη, τα οποία από μόνα του όχι μόνο δεν θα έβγαιναν από την ιστορία του κόσμου, θα ήταν σε πολύ δυσμενεί οικονομικέ συνθήκε. Πολλοί από εσά γνωρίζουν πώ ήσασταν πριν ενταχθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ξεχνάτε. Αυτό ισχύει για όλους και για τη χώρα μου που μπήκε πριν από πάρα πολύ καιρό, αλλά από αυτή τη σταδιακή διαδικασία συμμετοχής στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε να αποκομίσει πάρα μα πάρα πολλά ωφέλη. Και νομίζω ότι αυτό συνέβη για όλους μας. Δεν ήταν μόνο η διεύρυνση των αγορών, αλλά ήταν μια σειρά από σταδιακών κανόνων που μας επέτρεψαν να γίνουμε αυτή η οικονομική ε, δύναμη που είμαστε αυτή τη στιγμή. Εμείς τώρα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σίγουρα σεβόμενοι και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αλλά αυτό είναι ίδιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έγινε τίποτα χωρίς, όπως υπενθύμησε πριν ο, ο γερουσιαστής Μόντι, να ε, παραβιαστεί ουσιαστικά ο σεβασμός των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν μέσω του Συμβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εμείς υπενθυμίζουμε σε εσά, σε εσά σε αυτή την έκθεση, ότι θα πρέπει να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γκρινε εδώ δεν ωφελούν πρέπει να μπορέσετε να ζητήσετε από τι κυβερνήσει σα να λογοδοτήσουν. Τι πάνε να κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μιλήσετε μαζί του, να του δώσετε εντολέ. Υπάρχουν κοινοβούλια που δίνουν συγκεκριμένε εντολέ στι κυβερνήσει του όταν έρχονται στι Βρυξέλλε. Υπάρχουν άλλα βέβαια που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το ζήτημα και μετά απλώ φροντίζουν να διαμαρτυρηθούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για την κυβέρνησή του που δεν σεβάστηκε μια εντολή που δεν έλαβε και επομένω έκανε ό,τι ήθελε και ε, ίσως δεν τους αρέσει και δεν αρέσει και στους πολίτες μετά. Εμείς λοιπόν σας εκλυπαρούμε πέραν των πολιτικών σας θέσεων, από εκεί και προφανώς ο καθένας έχει τις πολιτικές του θέσεις. Όταν όμως συζητούμε για θεσμικά όργανα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχουν ε, οι πολίτες εδώ απ' έξω που διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται γιατί έχουμε κρίση και δεν έχουμε απαντήσει επαρκώς. Εδώ όμως αυτό που συζητάμε είναι πώς, και αυτή είναι μια συζήτηση θεσμική, όχι πολιτική, πώς μέσα από θεσμικές βελτιώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στις κείμενες συνθήκες, μπορούμε να έχουμε πιο δημοκρατικό διάφανο και σαφέστερο για τους πολίτες ε, το όλο σύστημα διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε μέσω μιας καλύτερης σχέσης μεταξύ ημών και εθνικών ε, κοινοβουλίων, μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και των εκπροσώπων τους να είναι πιο λειτουργικός ο συνολικός μηχανισμός μιας Ένωσης που δεν έχει μόνο 28 κράτα μέλη, αλλά και εντό των κρατών μελών μπορεί να έχει και περιφέρειες με νομοθετικές εξουσίες, ακόμα και κρατήδια με νομοθετικές εξουσίες. Αυτή η διαδικασία, δεδομένου λοιπόν ότι είναι σύνθετη, θα πρέπει να ρυθμιστεί, ε, να τη λαδώσουμε και μέσω θεσμικής διαδικασίας για να έχουμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα προφανώς και δεν προκύπτουν από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, όπως λένε οι Άγγλοι, δεδομένου ότι ακόμα έχουμε αγγλική καμπίνα εδώ, ε, να έχουμε deliver, να παραδίδουμε αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον συνάδελφο Μπροκ. Εάν λοιπόν έχετε χρόνο να σταθείτε λίγο περισσότερο στο ζήτημα και στα έγγραφα στα οποία σας υποβάλλουμε, ε, θα ήταν χρήσιμα και για σας, ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε πολύ καλύτερα στα κοινοβούλια σας αυτή την εργασία και κατά την ανωδική φάση, την ομοθετική, αλλά και στη φάση της εφαρμογής και της γνώσης. Κυρίως, όπως γνωρίζετε, οι χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι απαραίτητη, Καλύτερα λοιπόν να λειτουργήσει η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξημείνου και στις μεταξύ μας σχέσεις και για να γίνει αυτό πρέπει ε, να ε, προσπαθήσουμε να έχουμε στο τέλος τα αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι. Να σας ευχαριστήσω, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε και το γεγονός ότι συχνά η λειτουργία των θεσμών είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις πιο πολιτικές πτυχές που πολλοί από εσά έφυξαν σήμερα. Και πέραν αυτού είναι προφανές ότι και εντός της συνθήκης υπάρχουν κανόνες και για να προχωρήσουμε με διαφοροποιημένο τρόπο για όσους θέλουν να προχωρήσουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση μπορούν να το κάνουν και βάσει των συνθήκων. Αυτοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μπορούν κάλλιστα να το κάνουν και πάλι εντός της συνθήκης και η, η συνθήκη, όπως είναι γνωστό και μας το υποθύμησε και ο Άγγλος συνάδελφος, επιτρέπει και αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν πραγματικά θεωρεί κάποιος ότι δεν μπορεί να αντέξει την παραμονή του σε αυτή την Ένωση. Έχασα και τη φωνή μου, οπότε σταματάω. Ο Έλμαρτ, ε, σε ένα λεπτό να απαντήσει, να δώσουμε ένα λεπτό. Ναι, σας ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της ε, λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 κράτη-μέλη και οι αποφάσεις για την ενιαία αγορά λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία κανονικά. η δημιουργία της ε, αγοράς ήταν ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο θέμα, η κυριαρχία. Τα κράτη-μέλη, όπως είπα, κατέχουν τις αρμοδιότητες. Όταν όμως εκχωρούνται, ε, είναι μοιρασμένη η κυριαρχία και όταν λαμβάνεται σχετική απόφαση θα πρέπει να, να γνωρίζουμε τη σχετική απόφαση. Μπορεί κανείς να προσφυγεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί κανείς από μία απόφαση που ήδη έχει ληφθεί να απόσχει. δηλαδή να πάρει πίσω μία αρμοδιότητα την οποία ήδη έχει χωρίσει έτσι επειδή θέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να συνοψίσω και να κλείσουμε τη συζήτηση. Αναφερόμενοι σε ένα θέμα το οποίο έφυξαν πολύ. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και σκεφτούμε τους πολίτες σε αυτή τη συζήτηση φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι τα τελευταία χρόνια, μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες, οι κοινωνίες οι ευρωπαϊκές έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όσον αφορά την πρόσβασή τους στην πληροφορία έχουν αλλάξει τα πράγματα με λίγα λόγια. Αναφέρονται τα θέματα αυτά στην έκθεση. Επομένως το ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το περιθώριο ελιγμών που μας αυθύνουν οι συνθήκες για να προσερμόσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεσμικό της οικοδόμημα σε αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί στην κοινωνία. γιατί το ζήτημα αυτό απασχολεί και πρέπει να απασχολεί όχι μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και τα εθνικά, τους εθνικούς θεσμούς και στο εθνικό επίπεδο οι πολιτικοί θεσμοί έχουν αποτύχει συχνά να εκφράσουν τους πολίτες. Φαίνεται αυτό στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι νέοι. Πολλοί θεωρούν ότι αυτά, ε, τα, ε, αυτοί οι μηχανισμοί, αυτοί οι θεσμοί είναι μέρος του κατεστημένου, μας αντιμετωπίζουν με καχυποψία και θεωρούν ότι είμαστε παροχημένοι. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ένα ε, πρόβλημα μόνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και των εθνικών θεσμικών οργάνων. Επομένως, μια, ένα, μια εναλλακτική πρόταση, μια διαφορετική άποψη πρέπει να εκφραστεί όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Από την δικιά μας την πλευρά Πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πιέσει για να υιοθετηθούν προτάσεις και να βρεθούν λύσεις για θέματα που είναι σημαντικά για τους πολίτες. Έχουμε δημιουργήσει, για παράδειγμα, επιτροπές οι οποίες έχουν συζητήσει για το ζήτημα της ανισότητας, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς ή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων, να βελτιωθεί η λογοδοσία και αναρωτιέμαι, μπορούμε να βρούμε έναν απερκή αριθμό αντίστοιχων πρωτοβουλειών στο εθνικό επίπεδο. Εάν όχι και φοβάμαι πως όχι, πρέπει να συνεργαστούμε για να δοθούν τέτοιες απαντήσεις στους πολίτες και εθνικά. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια γενικό, ένα γενικότερο αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων. Και ο, πιστεύω και κοιτώ τον κύριο Σέπφιλτ που έχει ασχοληθεί με το θέμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πολύ, ε, τεράστιο λάθος όταν δεν ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλίε Ευρωπαίων πολιτών που είχαν αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο, το εργαλείο τη πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, είχαν συλλέξει μέχρι και ένα εκατομμύριο υπογραφέ και το ζήτημά του δεν ε, ε, ετέθη, δεν, το, δεν απάντησε καν σε αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το ίντερνετ, τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσουμε την διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ραμόν ε, το πρωί μας μίλησε για το ζήτημα αυτό και, και τη σύνδεσή του με την ηλεκτρονική δημοκρατία. Επίσης το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας το έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς στην Ευρώπη ούτε στο ευρωπαϊκό ούτε στο εθνικό επίπεδο. Και εδώ πιστεύω συμφωνούμε και βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει μια ανάγκη να αλλάξουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που, λειτουργούμε. Φαντάζομαι επίσης συμφωνούμε και σε αυτό που εξέφρασε ο κ. Μόντι και ο κ. Βιτορίνο, ότι πρέπει να έχουμε ε, να εστιαστούμε σε εκείνες τις πολιτικές που θα, θα αντιμετωπίσουν τα θέματα που κυρίως απασχολούν τους πολίτες, τους φόβους που κυρίως έχουν οι πολίτες. Και επίσης να μεταρρυθμίσουμε τους θεσμική μας λειτουργία έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν οι διάφοροι θεσμοί καλύτερα στις κρίσεις. Γιατί μας περιμένουν και άλλες κρίσεις στην Ευρώπη. Κλείνοντα θέλω να αναφερθώ και στη συνθήκη. Γιατί εκείνοι από εμά που σοβαρά σκέφτονται την πιθανότητα αναθεώρησης της συνθήκης, το προτείνουμε αυτό γιατί. Γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο η τρέχουσα συνθήκη περιγράφει την τρόπο διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη ξεπερασμένη. Δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν εξασφαλίζουν στους πολίτες ότι αν προσπαθήσουν να συμμετάσχουν θα έχουν κάποιο αντίκτυπο δεν εγγυάται η συνθήκη στους πολίτες που θα προσπαθήσουν να εκφράσουν την άποψή τους ότι θα εισακουστεί. Πρέπει λοιπόν να την επενεξετάσουμε τη συνθήκη υπ' αυτό το πρίσμα για να δούμε πώς μπορούμε να έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες μεγαλύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση στην ευρωπαϊκή ε, λήψη αποφάσεων. Και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να συσκεφθούμε για να καταλήξουμε σε ένα κοινό όραμα για το μέλλον και ρεαλιστικό αλλά και ε, κοιτώντας ε, μακριά. Γιατί έχουμε κοινέ αποφάσει δηλαδή κατά το παρελθόν και πρέπει να, πραγματικά να τι σεβαστούμε και να, να, να δεσμευτούμε ότι θα τι σεβόμαστε γιατί πιστεύω ότι εάν ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία, κάποιοι θα έρθουν μαζί μας, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσουμε στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, γιατί αυτό πιστεύω δεν θα ήταν επικοδομητικό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Όπως είχα και το πρωί, είχα πει και το πρωί, ε, θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξανασυναντηθούμε για να συζητηθήσουμε ε, την έκθεση εφαρμογής, δηλαδή την έκθεση που εξετάζει ε, τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην εφαρμογή των τρεχουσών συνθηκών για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνει γιατί ε, πιστεύω ότι χρειάζεται να πάμε ένα βήμα παραπέρα από τον πολιτικό, στον πολιτικό διάλογο. Να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι όλοι οι συνάδελφοί μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν εκφράσετε σχετικό ενδιαφέρον, με μεγάλη χαρά θα επισκεπτόντουσαν τις χώρες σας για να σας παρουσιάσουν τα θέματα που τους απασχολούν, τις εκθέσεις που προετοιμάζουν το γνωρίζετε, ε, θα ήθελα να το ε, επισημάνω για άλλη μια φορά ε, και να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επιθυμεί πάντα τη συνεργασία μαζί σας. Καλό απόγευμα αν μείνετε στις Βρυξέλλες, καλό ταξίδι αν γυρίζετε πίσω. λια τη συνεδρίαση τη κοινή συνεδρίαση των Εθνικών Κοινοβουλίων και τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ θα συνεχίσει τι εργασίε τη αμέσω μετά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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Так, так, короче. Thank you. Συνάδελφοι, μήπως μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα θυμάστε ότι το πρωί πριν την έναρξη της συνεδρίασης ε, της διακοινοβουλευτικής ε, ξεκινήσαμε τη συζήτηση της γνωμοδότησης ε, για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Σας παρουσίασα τα βασικά σημεία της γνωμοδότησης που εκπώνησα και το επόμενο στοιχείο αυτή τη συζήτηση είναι να ακούσουμε του σκιώδει εισηγητέ. Είναι παρούσα η Μερσέντε Μπρέζο. Θα τη δώσω λοιπόν το λόγο και κατόπιν θα σα ενημερώσω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση τη νομοδότηση αυτή. Μερσέντε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι για να επισέλθουμε τώρα σε λεπτομέρειες για μια τόσο περίπλοκη συζήτηση. Να σας δώσω και χρόνο να βάλετε τα ακουστικά σας. Γενικά μου φαίνεται ότι η εκθεσή σας είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιες συγκεκριμένε παρατηρήσεις. Ε, διότι αυτά τα οποία προτείνεται ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να τα δεχτούμε, τα συμμεριζόμαστε κι εμείς, εξετάζουμε αν λείπει τίποτα ε, και θα δούμε αν ε, θα πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες. Ε, προς το παρόν είμαστε ικανοποιημένοι από τις ε, προτάσεις σας. Δεν έχουμε βέβαια καταφέρει να τα δούμε, ε, αλλά μέχρι τις 7 του μηνός θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η πτυχή που αναφέρεται στις χώρες που σιγά σιγά εντάσσονται στο σύστημα να προβλέψουμε δηλαδή να έχουν κατάλληλη πρόσβαση ώστε να είναι καλύτερη μετάβαση. Ε, συμφωνούμε με αυτό. Ε, ε, κατά τα άλλα επιφυλασσόμεθα θα κάνουμε κάποια στιγμή κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τους Κιώδης εδώ. Θα ήθελα απλώ να σας ενημερώσω. Ε, κάνω έκκληση προς τους Κιώδης. Ε, αν καταθέσουν τροπολογίες θα πρέπει να σεβαστείτε την αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής μας. Ε, η Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι επί της ουσίας αρμόδια. προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 7η Δεκεμβρίου, υποθέτουμε, ε, στις 6 ώρα, Σεπτέμβριο Επιπρόεδρος. Θα ψηφίσουμε στις 30 Ιανουαρίου του 2017 εκτός και αν υπάρξει κάποια ριζοσπαστική αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ΕΚΟΝ ώστε ε, να είναι περιττό να πάμε εμεί τον Ιανουάριο για την ψηφοφορία. Προς το παρόν αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Πέρασε του, προγρα... σημείου αυτού και περνάμε στο τελευταίο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να το βρω, ελπίζω. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον δεν επέστρεψε. Ε, τα θυμάμαι βέβαια αυτά που μου είπε. Α, είστε εδώ, συγγνώμη. Πρέπει να βγάλω και τα γυαλιά μου να σας δω. Στο σημείο 7 έχουμε πρόταση τροποποίηση τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία, τη συνεργασία στα θέματα υπολογισμού και ε, στην υγιή ε, οικονομική διαχείριση. Ε, παραπέμφθηκε στην Επιτροπή μας γιατί υπήρχε ε, η υποψία ότι μπορεί να χρειαστεί αναθεώρηση των διαπραγματεύσεων για τη Διοργανική Συμφωνία και να καθοριστούν ε, να αναφερθούμε στο αποθεματικό για ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω το λόγο να μας εξηγήσετε κατά πάσα πιθανότητα ε, θα αναβάλουμε τις συζητήσεις λόγω των πληροφοριών που θα ακούσετε, αλλά θα αποφασίσετε στη συνέχεια. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η πρόταση τροποποίησης της Διοργανικής Συμφωνίας είχε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για το, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αποθεματικού Κρίσης. Ε, προχώρησαν τώρα τα πράγματα. Ε, πλησιάζουμε στην πολιτική συμφωνία και στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Ε, το Ευρωπαϊκό Αποθεματικό Κρίσης αυτή τη στιγμή δεν είναι τμήμα της συνολικής πολιτικής συμφωνίας από πλευράς ε, Συμβουλίου. Ε, έχουν βρει άλλο τρόπο να εγκρίνουν και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ευελιξίας που χρειάζονται, που σημαίνει ότι η τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας δεν χρειάζεται. Αυτή λοιπόν ε, η αλλαγή θα ε, προκύψει από το νομοθετικό πακέτο και ο κανονισμός για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα είναι το μέσο το οποίο θα μας οδηγήσει, βοηθήσει να το μετατρέψουμε σε νομικό κείμενο. Επομένως η τροποποίηση θα είναι περιττή κατά την απόψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής. Δεν θέλω να το κλείσω ακόμα γιατί υπάρχει μια επιρροελάχιστη περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει διοργανική συμφωνία, αναθεώρηση και δεν θα χρειαστεί αποθεματικό κρίτης. Ε, θα αλλάξουμε λοιπόν τα πράγματα. Σας ενημερώνω ότι προς το παρόν λοιπόν αναβάλλεται η απόφαση, αλλά θα το δούμε αυτό σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτό ήταν το τελευταίο ουσιαστικό σημείο. Στα διάφορα δεν έχω κάτι εγώ. Η επόμενη συνεδρίαση δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε γιατί δεν έχει καμία ουσία. Αν χρειαστεί θα το συζητήσουμε. Τελευταίο σημείο λοιπόν, ενημέρωση. Θα γίνουν δύο συνεδριάσεις πολύ σύντομα. Η 5η Δεκεμβρίου είναι η τακτική μας συνεδρίαση και 8 Δεκεμβρίου έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση και τις δύο στις Βρυξέλλες. Στις 8 του μηνός θα ψηφίσουμε τις δύο εκθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η συνεδρίαση αυτή. Γράφετε κάτι για μένα. Πες το. Α, και υπάρχει και η πρόταση που από ό,τι κατάλαβα έχει ήδη σταλεί στους συντονιστές. Μπορεί να γίνει συνεδρίαση των συντονιστών τη Δευτέρα στις 2 η ώρα. Γιατί η Δευτέρα είναι 5 του μηνός που συνεδριάζουμε στις 3. Αν μπορείτε να έρθετε νωρίτερα, αλλιώς ε, μετά τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι εγώ στις 2 προσγειώνομαι. Είναι λίγο νωρίς για μένα. Δεν έχετε διοικητικό αεροπλάνο ακόμα. Το προσπαθώ, το προσπαθώ έχει ένα ε, μεγάλο ελικόπτερο, δεν τα λέω όμως. Είναι και αυτά τα καρακάλα, τα ελικόπτερα που δεν αγοράζει η Πολωνία. Άμα θέλετε έχουν οι πολλά λοιπόν. Μήπως μου δανείσετε ένα, ε, θα μου ήταν χρήσιμο. Μετά προτιμάτε δηλαδή. Ναι, προτιμώ μετά. Και εσείς. Ναι, και εγώ το προτιμώ, γιατί έχω μια συνεδρίαση δύο αιών, ε, ωρών δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τελειώσω. Θα είναι μια συζήτηση γύρω στο μεσημέρι. Ορισμένε φορέ όμω είναι δύσκολο να φύγω ακριβώ στι δύο. Καλύτερα αργότερα λοιπόν, γιατί μπορεί να μην προλάβω. Λοιπόν, θα γίνει μετά λοιπόν τη συνεδρίαση. 6,5 ώρα θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ στι 5 Δεκεμβρίου. Τέλεια. Αν η συνεδρία τελειώσει νωρίτερα βεβαίω, θα συνεδριάσουμε νωρίτερα. Ευχαριστώ. Πέρασε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ σε όλου. Γεια σας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, μεταφραστές κλπ.